Okay. Welcome. Καλώς ήρθατε. Θα αρχίσουμε, διότι υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Καταρχήν, θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνεται. Και τώρα ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τον Τρίλογο. Ο πρώτος τρίλογος ε, ε, έλαβε χώρα στις 16 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Ε, σημειώθηκε πρόοδο και για πρώτη φορά συζητήθηκαν όλες οι ημερομηνίες οι οποίες θα καθοριστούν στο κείμενο. Υπάρχουν λοιπόν ελάχιστα εκρεμή. Η Κομισιόν λοιπόν ανέλαβε να κάνει δύο δηλώσεις, ένα για τις επιστροφές και, και μία δήλωση για τις πληρωμές και τέλος ο τρίλογος ελπίζουμε ότι θα είναι επαρκής για να ολοκληρωθεί το κίνημα μέχρι τις 29 Νοεμβρίου. Σχετικά με τις ε, ε, καταθέσεις, εγγύσεις καταθέσεων. Ε, ο πρώτος τρίλογος έγινε την πρώτη εβδομάδα στις 16 του μηνός στο Στρασβούργο. Το Συμβούλιο ανέλαβε την υποχρέωση για συνέχιση των διαβουλεύσεων. Επίσης αποφασίστηκε να ανοίξουν οι συζητήσεις στα τεχνικά θέματα. Ε, συζητήθηκε ένας κατάλογος τεχνικών θεμάτων με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προωθήθηκε στο Συμβούλιο και την Κομισιόν. Περαιτέρω συνεδριάσεις σε επίπεδο τεχνικό θα καθοριστούν. Σχετικά με το Μύθιτ. Ε, ο, καθη, ο εισηγητής κύριος Θέρμπερ ε, ξεκίνησε, μάλλον ε, μοίρασε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το Μύθιντ. Και τα σχόλια από τους σκιώδεις υπάρχουν σε αυτό το ερωτηματολόγιο. Θα τα βρείτε στο διαδίκτυο. Όλες οι πλευρές καλούνται να σχολιάσουν και όχι μόνο τα μέλη αλλά και οποιοδήποτε. Παρακαλώ να αντιδράσετε στη Γραμματεία έως τις 13 Ιανουαρίου 2012 και οι απαντήσεις αυτές θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη που ασχολούνται με την επανεξέταση του ΜΥΘΙΤ. Επίσης υπάρχει μια δημόσια ακρόαση στις 5 Δεκεμβρίου στο ε, ΜΥΘΙΤ και οι λεπτομέρειες και ο κατάλογος θα κυκλοφορήσουν το ταχύτερο δυνατό μόλις είναι διαθέσιμα. Επίσης θα ήθελα να πω στα μέλη ότι στην απογευματινή μας συνεδρίαση της 3ης 29 Νοεμβρίου θα ακυρωθεί διότι και όλα όσα έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της πρωινή συνεδρίασης. Το σχέδιο ημερησίας διατάξεως θα κυκλοφορήσει το συντομότερο. Και αυτό ε, σημαίνει ότι ενδεχομένως θα υπάρχει τριμερής διάλογος το απόγευμα. Και έτσι θα είναι ε, διαθέσιμοι επιθυμούντες να συμμετάσχουν. Αυτές είναι λοιπόν οι ανακοινώσεις και τώρα με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Επίτροπο κύριο Αλμούνια στην Επιτροπή για μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον ανταγωνισμό. Το θέμα αυτό το συζητήσαμε στις 22 Σεπτεμβρίου τελευταία φορά και βεβαίω προσβλέπουμε και στον καθορισμό μια ημερομηνία στο προσεχές έτος. Πάντως θα δώσω καταρχήν το λόγο στον Επίτροπο, ο οποίο θα μα ενημερώσει επί των θεμάτων των σχετικών με τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση που αφορά τον ανταγωνισμό περιλαμβανομένου και του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012. Και βεβαίως θα σας δοθεί ευκαιρία να απαντήσετε σε ερωτήσεις που ενδεχομένως θα θέσετε. Και θα σας δώσω τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού. Όταν λοιπόν μου ζητήθηκε από τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλω κάποιες ε, ιδέες για πρωτοβουλίες για το προσεχές έτος, σκέφτηκα ότι όλες οι πρωτοβουλίες που θα υιοθετηθούν θα πρέπει να συνδέονται με την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ανακτηθεί ένας βιώσιμος δρόμος προς την ανάπτυξη. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι πάντοτε σημαντική ώστε να διατηρείται η ενιαία αγορά όσο γίνεται πιο ανοιχτή, χωρίς εμπόδια, χωρίς προσκόμματα, με ελεύθερο ανταγωνισμό για όλους τους μετέχοντες και χωρίς στρεβλώσεις. Αλλά στις δύσκολες αυτές εποχές νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό η πολιτική ανταγωνισμού ως ένα θεμελιώδες μέσο διεύρυνσης ανοίγματο της αγοράς ώστε να δώσουμε νέα όθηση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και να βοηθήσουμε τις εταιρείες μας και ιδιαίτερως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως επίσης να δώσουμε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πολιτική ανταγωνισμού σε τέτοιες εποχές κρίσης ιδιαιτέρως είναι ε, το καλύτερο τόνοτικο για τις επιχειρήσεις. Προάγει την αποτελεσματικότητα, προετοιμάζει τις επιχειρήσεις για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και ενθαρρύνει την καινοτομία. Είναι αληθές ότι σε πολλούς τομείς, ε, και το γνωρίζετε αυτό επαρκώς, διότι ε, το φόρτος εργασίας σας αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια και το γνωρίζετε, τα ρυθμιστικά μέτρα είναι ζωτική σημασία για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αλλά η πολιτική ανταγωνισμού είναι θεμελιώδης ε, ακριβώς επειδή μέσω κυρώσεων μπορεί και εμποδίζει τα προσκόμματα εκείνα τα οποία διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας έγερσης ενός τείχους προστατευτισμού στις αγορές. Αυτά τα μέσα προστατευτισμού ή τα εμπόδια ε, προστατευτισμού είναι αν θέλετε μία προσπάθεια που γίνεται σε τέτοιες δύσκολες εποχές. Άρα λοιπόν, ε, ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις κάνουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν αφενός τους πελάτες τους και να διατηρήσουν το επίπεδο της επιχειρηματικότητάς τους. Έτσι λοιπόν, ε, έχω την πρόθεση να παρουσιάσω στους συναδέλφους μου την Κομισιόν μια πρόταση για κρατική βοήθεια και επίσης μια νομοθετική πρωτοβουλία για ενίσχυση ε, του ανταγωνισμού στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά πριν σας αναπτύξω περισσότερο τα δύο αυτά σημεία, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και ιδιωτέρω αυτή την Επιτροπή για τον επικοδομητικό διάλογο για την αναθεώρηση των κανόνων για τις κανόνων σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα μετά από μια μακρά περίοδο διαβουλεύσεων, κάτι το οποίο θα υιοθετηθεί από το Κολέγιο των Επιτρόπων τον επόμενο μήνα, το Δεκέμβριο. Το πακέτο λοιπόν μεταρρυθμίσεων βρίσκεται στην τελευταία ε, φάση σύνταξης. Έλαβα υπόψη πάρα πολλά σχόλια τα οποία ε, διατυπώθηκαν στην τελευταία δημόσια διαβούλευση. Έδωσα ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεση Σάιμον και τη συζήτηση γύρω από την έκθεση αυτή που έλαβε χώρα πρόσφατα, είμαι ακόμα ανοιχτός να τροποποιήσω κάποιες πτυχές των αρχικών μας προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήματα που διατυπώνονται και ιδιαίτερος θα πρέπει να ολοκληρώσω, να τελειοποιήσω την πρόταση για τα κατώτατα όρια του κανόνα de minimis, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχόλια που διατυπώθηκαν και συμφωνώ απολύτως με την έκθεση του Κοινοβουλίου για την ανάγκη κάλυψης περισσότερων κοινωνικών υπηρεσιών ε, σε σχέση με το πακέτο 2005 και τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενημέρωσης. Και πέραν αυτού, και τώρα αναφέρομαι στην πρώτη τροπολογία, ε, στην πρώτη πρωτοβουλία, συγγνώμη, θα καταβληθούν δηλαδή προσπάθειες εξορθολογισμού και ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Και με την έννοια αυτή, το προσεχές έτος θα δρομολογήσω μια νέα πρωτοβουλία, ούτως ώστε να είναι πιο σαφής η δική μας συνεισφορά στις κρατικές ενισχύσεις και επίσης στις στρατηγικές ε, δημοσιονομικού εξορθολογισμού που εφαρμόζονται στις χώρες μέλη. Θα ανοίξουμε τη συζήτηση ώστε να δούμε πώς η κρατική ενίσχυση μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη, στην καινοτομία, στις οικονομίες μας, στην ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να είμαστε αυστηρότεροι στους ελέγχους των κρατικών ενισχύσεων που μπορούν να διακυβεύσουν την, τους στόχους δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόζονται σχεδόν σε όλες τις χώρες μέλη ε, τα προσεχή χρόνια. Και ταυτόχρονα, όπως ακριβώς έκανα και με το πακέτο AGI, θα επιδιώξουμε να έχουμε αποτελεσματικότερες και πιο αποτελεσματικότερες και απλούστερες διαδικασίες. Αυτά λοιπόν θα συζητήσω μαζί σας πάντοτε. Σα... Είμαι ανοιχτό σε έναν ευρύ διάλογο, τον ευρύτερο δυνατό θα έλεγα. Και θα ήθελα να ακούσω τη δική σας συνεισφορά και απόψεις στη συζήτηση αυτή. Ούτως ώστε κατά το δεύτερο μέρος της εντολής μου ε, ως Επιτρόπου Ανταγωνισμού να αναπτύξω νέες πρωτοβουλίες λαμβάνοντας υπόψη ευρύτερες στρατηγικές, ευρύτερες προοπτικές. Έτσι λοιπόν η άλλη τώρα πρωτοβουλία για το 2012 αφορά το δικαίωμα των ατόμων και των επιχειρήσεων να, ε, να απαιτούν αποζημιώσεις όταν γίνονται παραβιάσεις της νομοθεσίας αντιτράστα. Έτσι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να απαλείψουμε όλα τα προσκόμματα και τα εμπόδια που υπάρχουν για την καταβολή αυτών των αποζημιώσεων. Επίσης θέλουμε να εισαγάγουμε μια εναρμόνιση, ιδιαίτερως μετά την απόφαση τη Φράιντερερ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που δείχνει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να προστατεύσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται, αλλά επίσης να δίδονται, να δίδεται και το δικαίωμα, να προστατεύεται μάλλον το δικαίωμα για αποζημίωση των ατόμων αλλά και των επιχειρήσεων. Όπως γνωρίζετε, αυτή η πολιτική η ιδιω, εφαρμογής ε, απαιτεί να υπάρξει δημόσια διαβούλευση παράλληλα με όσα έγιναν τους προηγούμενες μήνες. Και βεβαίως αν χρειάζεται να υπάρξουν συλλογικές δράσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατές με τις αρχές που έχουμε υιοθετήσει στην οριζόντια προσέγγιση μας για την συλλογική αποκατάσταση. Λοιπόν, ε, καταρχήν, πριν από το τέλος αυτού του έτους θα υιοθετήσουμε την απόφαση να παρατείνουμε και στο προσεχές έτος την εφαρμογή των ειδικών κανόνων κρίσης για κρατικές ενισχύσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Όπως γνωρίζετε, πρόθεσή μου ήταν να ακυρώσω, να σταματήσω αυτό το καθεστώς της κρίσης στο τέλος αυτού του έτους. Αλλά επειδή η κατάσταση στην αγορά δεν είναι επαρκής, θα παρατείνουμε το καθεστώς αυτό για το προσεχές έτος, έως ότου οι συνθήκες της αγοράς εξομαλυνθούν. Και με την παράταση αυτή και μάλλον στο πλαίσιο της παράτασης αυτής θα προσαρμόσουμε τις τιμές των κρατικών εγγυήσεων λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που προέκυψαν τα τελευταία τρία χρόνια από τη στιγμή δηλαδή που υιοθετήσαμε ε, την πρώτη απόφαση για τα όρια, το ύψος των κρατικών εγγύσεων. Και επίσης θα εξηγήσουμε υπό ποιες συνθήκες θα γίνονται οι ενισχύσεις των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, διότι όπως αποφασίστηκε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο, αυτή είναι η στόχη για ενίσχυση κεφαλαϊκή των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων. Αλλά σε περιπτώσεις που το ιδιωτικά κεφάλαια δεν είναι διαθέσιμα, δημόσια κεφάλαια μπορούν να διατεθούν και στην περίπτωση αυτή πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογουμένων που θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιοποίηση των ε, χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή ούτως ώστε να διασωθούν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Μόλις λοιπόν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς θα εισαγάγουμε ένα νέο καθεστώς για φυσιολογικές ε, συνθήκες ενίσχυσης των χρηματοοικονομικών ε, Ιδρυμάτων. Και με τον ίδιο τρόπο, τον, το προσεχή Οκτώβριο, θα υιοθετήσουμε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για μη χρηματοοικονομικά ιδρύματα, που και αυτό θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω ότι ετοιμάζουμε νέες κατευθυντήριες γραμμές που θα υιοθετηθούν το 2012 στον τομέα της ε, των αεροπορικών γραμμών, ε, δηλαδή αεροπορικές εταιρείες και υποδομές αεροδρομίων, νέες κατευθυντήριες γραμμές για την αυσιπλοεία και η δημόσια διαβούλευση θα ξεκινήσει πριν το τέλος αυτού του έτους. Θα ενημερωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για risk capitals. Θα προσδιοριστούν οι νέες στρατηγικές. Θα υιοθετήσουμε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ε, περιφερειακή ανάπτυξη, έρευνα και καινοτομία. Μέχρι το τέλος του 2012 θα επανεξετάσουμε την ανακοίνωση κρατικών ενισχύσεων για ε, πιστώσεις εξαγωγών και ασφαλιών κατευθυντήριες ε, γραμμές για τον κινηματογράφο και κρατικές ενισχύσεις δηλαδή ε, σε αυτό το τομέα που και επίσης θα υιοθετηθούν στο τέλος του 2012. Και τέλος, στις αρχές του 2012, το πρώτο τέταρτο, θα υιοθετήσουμε κατευθυντήριες γραμμές για κρατικές ενισχύσεις που θα βοηθήσουν τον κλάδο τον ενεργειακό και ιδιαίτερος αυτούς που εκπέμπουν διοξίδιο του ε, άνθρακα. Ε, διότι θέλουμε να, να ενισχύσουμε ακριβώς αυτούς τους φορείς και θέλουμε να περιορίσουμε την διαρροή άνθρακα και επειδή η, τιμή του, του ηλεκτρικού ρεύματος ε, είναι πολύ ψηλή υπό αυτές τις συνθήκες, ταυτόχρονα η αποζημίωση μπορεί να είναι υψηλή, ούτως ώστε να στείλουμε και το κατάλληλο μήνυμα στο, στους παραγωγούς. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι έχουμε διαβουλεύσεις με τις χώρες μέλη, με τους ε, κλάδους και προτίθεμε να υιοθετήσω αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2012. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος και τώρα παρακαλώ ερωτήσεις ε, οι οποίες υποβάλλονται ελεύθερα. Λέω τα ονόματα. Anybody else? Ωραία, λοιπόν. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας. Ε, θα υποβάλλετε την ερώτηση και θα απαντάει ο Επίτροπος καταρχήν σε κάθε ερώτηση. Αν είστε σύντομοι, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αν ε, τελικώς ε, δεν μπορέσουμε, θα θέσω περιθώριο χρόνου. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, τις ε, για την εισήγησή του. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για, το... για του χρόνου, για την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ήθελα ορισμένες ε, πληροφορίες για ορισμένες πτυχές των θεμάτων. Για παράδειγμα, στα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, ποιες είναι οι αντισταθμίσεις που προβλέπονται. Γιατί έχουμε μία σειρά αντισταθμίσεων που ακούσαμε με βάση τις ανάγκες του εκτελεστικού, έτσι ώστε να έχουμε συστήματα αρρωγής ή εγγύησεων. Νομίζω ότι η εγγυσεων νομιζω οτι η επιτροπη θα πρέπει να δράσει σαφώς ως προς αυτές τις πτυχές. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω πώς κρίνεται τις πιστοτικές ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς ε, αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό ως προς τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ε, πρωτοβουλία της Κομισιόν για μη... και από ό,τι ακούσαμε θα γίνει μείωση της βαθμολόγησης της Γαλλίας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να μας δώσετε ε, στοιχεία. Πώς όλα αυτά συνάδουν με την πολιτική ανταγωνισμού και μπορεί να υπάρξει στρέβλωση ανάλογα με τη λειτουργία των αγορών. Και τέλος, ως προς τον τομέα της ναυπηγικής, νομίζω ότι χρειάζεται, χρήση βοηθείας. Υπάρχουν προβλέψεις. Μου είπε η πρόεδρος να μην μακρηγορώ. Να απαντήσω, να απαντήσω. Θα ήθελα να απαντήσω στο φίλο μου τον Αντολίν. Ε, τηλεγραφικά. Ως προς τα πριμ, των τραπεζών που, έχουν, που λαμβάνουν κρατική επιδότηση. Επειδή ελέγχουμε τις κρατικές επιδοτήσεις, μπορούμε να επιβάλλουμε λύσεις έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο είναι συμβατή η βοήθεια αυτή, η επιδότηση αυτή, ανάλογα με τα ενδεχόμενα κέρδη, τη στιγμή που μιλάμε για δημόσιους οργανισμούς και υπάρχει περίπτωση περιορισμού των μερισμάτων. και κατά πόσο μπορούν να καταβληθούν τα κούπονς σε περίπτωση ε, σταθερής απόδοσης, καθώς και άλλα μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει σωστή κατανομή των ε, προσπαθειών αυτών. Δηλαδή, από νομικής πλευράς δεν μπορούμε να απαγορέψουμε αυτό το ε, είδος της αντιστάθμισης. Ο συνάδελφός μου, ο Μισελ Μπαρνιέ, που θα έρθει σήμερα το απόγευμα εδώ, θα προπαρασκευάσει μία πρόταση νομικού πλαισίου, νομικού περιεχομένου, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να ε, ελέγξουν την κατάσταση, διότι τα κράτη το που προβαίνει στην ε, κρατική επιδότηση να μπορεί να την χορηγήσει υπό όρους. Αυτό το βλέπουμε και στην ε, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή υπάρχει ε, ένα όριο 50% ως προς τα πριμ αυτά. Αλλά δεν μπορούμε προς το παρόν, δεν υπάρχει ε, μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Ως προς τη ροή κονδυλίων, και εδώ δεν υπάρχει όριο. Δηλαδή, μία χρηματοοικονομική αρχή θα πρέπει να τηρεί τις ε, βασικές τις, ε, τα βασικά τις, τις βασικές δεσμεύσεις, δηλαδή να χρηματοδοτεί ανάλογα με τις οικονομικές ανάγκες. Εμείς προσπαθούμε να ορίσουμε αυτές τις ε, κεφαλαιακές ροές ανάλογα με τις, με τις κρατικές ή δημόσιες δεσμεύσεις. Γιατί θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτές οι δεσμεύσεις από τις χρηματοοικονομικές αρχές. Με βάση της πρόσφατης συμφωνία στο ΕΚΟΦΗΝ, που υποστηρίχθηκε και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ε, εκ νέου κεφαλαιοποίηση των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, τη στιγμή που προβλέπεται αυτό από τις κρατικές αρχές ορίζουμε τους όρους αυτής της ε, εκ νέου κεφαλαιοποίησης και στη συνέχεια οι εποπτικές τραπεζικές αρχές θα πρέπει να δουν μέχρι ποιού σημείου πληρούνται οι όροι με βάση τις κεφαλαιακές αλλαγές τύπου Cortier 1 μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, εκ νέου κεφαλαιοποίησης που ορίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες ενεργητικού τύπου Tier 1. Ως προς τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, επαναλαμβάνω αυτά που είχα πει εκ των προτέρων. Το πρόβλημα αυτών των οίκων αξιολόγησης δεν είναι προβλήματα τύπου αντιτράστα. Υπάρχουν άλλα προβλήματα ευρύτερης εμβέλειας και ο κανονισμός που εγκρίναμε τις προηγούμενες μέρες αφορά την αντιμετώπιση συγκεκριμένων, συγκεκριμένων μάλλον σύγκρουση συμφερόντων τέτοιων προβλημάτων και όχι τύπου αντιτράστα. Και ως προς τις καταχρήσεις, με την αποστολή πληροφοριών συγκεκριμένου τύπου σε χρηματοπιστωτικούς φορείς, πριν δοθούν αυτές οι πληροφορίες στην αγορά, κάτι το οποίο μπορεί να έγινε στη Γαλλία, αυτό είναι κάτι που έχει σχέση με τις ε, καταχρήσεις της αγοράς και θέμα χρηματοοικονομικής πειθαρχία. Δηλαδή δεν έχει σχέση με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές που εφαρμόζουν οδηγίες ως προς τον τομέα της ναυπηγικής. Εμείς ορίζουμε νέες κατευθυντήριες γραμμές δίδουμε, προσδίδουμε μεγάλη σημασία στον τομέα της ναυπηγικής. Βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας διαβουλεύσεων. Αν σας ενδιαφέρει το θέμα, μπορώ να προσέλθω εδώ και να σας το επεξηγήσω. Και αυτό το βλέπουμε μαζί με τον τομέα του άνθρακα. Εγώ ορίζω αυτές τις ειδικέ κατευθυντήριες γραμμές, όχι δηλαδή οριζόντιου τύπου, αλλά εγκαρσίου, για να δούμε πώς μπορεί να αναδιαρθρωθεί ο τομέας. Ο τομέας της ναυπηγικής αντιμετωπίζει δυσκολίες, υπάρχουν ιδιαιτερότητες του τομέα αλλά και εκεί ισχύουν οι γενικές αρχές, δηλαδή οι κρατικές ενισχύσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κρατήσουμε τεχνητά εν ζωή έναν τομέα ή ένα φορέα ο οποίος είναι εθνησίγενης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι ενισχύσεις επιτρέπονται για αυτό το τομέα, για να είναι ανταγωνιστικός, για να καινοτομήσει, και τι ενισχύσεις επιτρέπονται. Γιατί το δημόσιο χρήμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρατήσουμε εν ζωή έναν τομέα ο οποίος δεν είναι βιώσιμος. Δεν μπορούμε τεχνητά να κρατάμε στη ζωή έναν ασθενή ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να επιζήσει. Έχουμε μία ώρα, δέκα ερωτήσεις, δώδεκα έξι λεπτά, τώρα περνάμε στα δώδεκα. Λοιπόν, τώρα θα σας βλέπουμε σε διάδες. Η Βάρη και μετά η Σόφη. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Επιτρόπε, θα ήθελα να σα ρωτήσω για την ε, κοινή γεωργική πολιτική. Δεν μπορείτε να μιλήσετε φιλανδικά σήμερα, δυστυχώ. <laughs> Ετε. Κασ. Μην το tõlge λέμε. Λοιπόν, κύριε Επίτροπε, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για την ε, κοινή γεωργική πολιτική. Καταλαβαίνω βεβαίω πως ε, δεν είναι η δική σας ε, αρμοδιότητα, αλλά μια που μιλάμε για το 40% του προπολογισμού, και 100% της ε, αεροτρέας γης νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα και γνωρίζουμε βεβαίως ποιο είναι το όραμα του Επιτρόπου Γεωργίας για το μέλλον της Γεωργίας μιλάμε εκεί πέρα για τις άμεσες ε, πληρωμές και για την μεταβατική περίοδο ε, στην οποία όλα τα κράτη-μέλη θα λαμβάνουν μια μέση πληρωμή στρέμμα και βεβαίως ε, η μεταβατική περίοδος είναι 17 ολόκληρα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν πως υπάρχει μία κάποια στρέβλωση εδώ πέρα. Εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει μία άμεση μετάβαση, να, πρέπει να καταργήσουμε τι άμεσε πληρωμές. Δεν ξέρω. Να πάνε τα λεφτά στη διαστημική έρευνα. Τι άποψη έχετε από αυτό. Λοιπόν, Σόφη, τώρα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Επίτροπε. Δύο σύντομες ερωτήσεις, μία πιο γενική. Έχω την αίσθηση πως η γενική αυτή συζήτηση περί κρατικών ενισχύσεων η ε, έννοια της μείωσης των κρατικών ενισχύσεων ε, έχει χαθεί γιατί υποτίθεται πως η αρχή είναι πως δεν επιτρέπονται και μετά υπάρχουν διάφορες εξαιρέσεις αλλά κατ' ουσίαν μιλάμε για αναδιανομή ε, κρατικών ενισχύσεων παρά για μείωσή τους. Ναι εντάξει αναφέρατε τον τίτλο της συζήτησης ο οποίο είναι πώ μπορεί να συνεισφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις στην ανάπτυξη και μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά ταυτόχρονα στρεβλώνεται ο ανταγωνισμό και μιλάμε για δημόσιο χρήμα σε καιρού λιτότητα. Και έχω την αίσθηση καμία φορά πως η ήπειρο μα ε, εθίζεται στις επιδοτήσεις και εγώ θα ήθελα να συζητηθεί το πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτή την εξάρτηση από τις επιδοτήσεις αντί για να την αυξήσουμε. Το δεύτερο ερώτημα είναι πιο συγκεκριμένο. Σήμερα η κυβέρνηση της ε, Ολλανδίας μάλλον θα αντιμετωπίσει ε, ψήφο δυσπιστίας ε, και το ζήτημα είναι, το πιστεύετε είτε όχι, οι κρατικές ενισχύσεις στην κοινωνική στέγη. Νομίζω λοιπόν πως πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο η συζήτηση στην Ολλανδία και θα ήθελα από σας κάποιες διευκρινήσεις. Γιατί κάποια κόμματα υποστηρίζουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε υποχρεωτικό κατόφλι στον, ε, στην κοινωνική στις εργατικέ κατοικίε στην ε, Ολλανδία. Εγώ θεωρώ πώ αυτό δεν ισχύει. Θεωρώ πώ ε, αυτό το αποφάσισε η Ολλανδική κυβέρνηση. Και η Κομισιόν απλά λέει αν ισχύουν οι κανόνε. Από την άλλη, μα λέει η κυβέρνηση πώ θα αλλάξουν οι κανόνε των κρατικών ισχύσεων και τότε θα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Ολλανδία. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Α, δεν ξέρω, μπορεί να μην είμαι ενημερωμένη. Ε, αν μπορείτε να μα βοηθήσετε. Και τέλο, θα ήθελα να μάθω Εάν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να υπάρχει μια επίσημη κανταγγελία από τους εργολάβους ε, στην Ολλανδία για το τι μπορεί να θεωρηθεί κοινωνική παροχή στέγασης και το τι είναι εμπορική δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ. Για το ερώτημα του φίλου μου του κυρίου Πάνταρ. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να απαντήσω στο ερώτημά σας. Δεν είμαι ειδικό στην κοινωνική πολιτική. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι πως οι αποφάσεις ε, της Κομισιόν Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για την κοινωνική πολιτική εξορισμού δεν μπορούν να παραβαίνουν τους κανόνες μας. Γιατί είναι οι κανόνες. Οπότε όλες οι αποφάσεις για πληρωμές ε, που έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση εξορισμού δεν ε, μπορούν να θεωρηθούν ε, κρατική ενίσχυση. Επί της ουσίας τώρα, το ερωτήματό σας αντιλαμβάνομαι τη, τη σημασία του, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν, δεν είναι ο τομέας μου. Είμαι περισσότερο στα αστικά παρά στα της υπαίθρου. Τώρα για τη μείωση ή την αύξηση της κρατικής ενίσχυσης. Δεν είναι αυτό δική μας απόφαση, είναι απόφαση των κρατών μελών. Υπάρχουν κράτη-μέλη με πολλές ε, κρατικές ενισχύσεις στον προϋπολογισμό τους, στο πρόγραμμά τους, ε, αρκεί πάντα να είναι συμβατή με τις καθητήριες γραμμές. Κάθε φορά που δεν είναι συμβατή ε, έχουμε αρνητικές αποφάσεις με ανάκτηση, αν ε, χρειαστεί. Αλλά τώρα, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να αυξηθεί ε, το ύψος ε, των δημοσίων ενισχύσεων δεν είναι απόφαση της Κομισιόν. Εμείς απλά βλέπουμε αν είναι συμβατή ή όχι η ενίσχυση ή αν είναι κάτω από τον κανόνα του επιέλατον δεν θεωρείται ενίσχυση. Δεδομένου του ότι είμαστε σε μία περίοδο η οποία θα διαρκέσει κάποια χρόνια ε, φιλόδοξης ε, δημοσιονομικής ε, εξυγίανσης στα περισσότερα κράτη-μέλη θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο εστιασμένοι στο πού είναι ασύμβατες κρατικές ενισχύσεις και πού δεν θα πρέπει να σπαταλάμε δημόσιο χρήμα και που δημιουργεί επίσης ε, στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Βεβαίως, το σκεπτικό είναι να αποφύγουμε ακριβώς ε, στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Αλλιώς, γιατί να ελέγξουμε. Γι' αυτό ακριβώς ελέγχουμε τις ε, δημόσιες ενισχύσεις. Αλλά όπως σας είπα, σε καιρό λιτότητας, όταν θα πρέπει να ενισχύσουμε το δυναμικό της ανάπτυξης, πρέπει να είμαστε πιο εστιασμένοι και να επικεντρωθούμε στο να χρησιμοποιούμε τα, το δημόσιο χρήμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, εκεί όπου μπορεί να αυξηθεί η ανάπτυξη και να είμαστε αυστηρότεροι στους τομείς όπου η χρήση του δημοσίου χρώματος όχι μόνο στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, αλλά είναι και σπατάλη. Αυτές είναι οι αρχές μου. Και από όταν ξεκινήσαμε εμείς ε, να εισάγουμε την οικονομική ανάλυση στις κατευθυντήριες γραμμές μας, νομίζω πως βελτιώνουμε την ε, αποτελεσματικότητα των ελέγχων μας, που δεν έχει μόνο στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, αλλά προσπαθούμε να δούμε πώς χρησιμοποιούνται καλύτερα τα δημόσια αυτά κονδύλια. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας και η φιλοσοφία της Κομισιόν. Τώρα, για την κοινωνική στέγαση τις εργατικές κατοικίες. Το έχω πει πολλές φορές σε δημόσιες και σε διμερείς συναντήσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Δεν είμαι Ολλανδός πολιτικός και ποτέ δεν θα γίνω Ολλανδός πολιτικός. Ε, δεν ξέρω, μπορεί στο μέλλον. Α, δεν το νομίζω. Οπότε δεν ε, έχω εμπλακεί εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Ξέρω πως είναι πολύ σημαντική στην Ολλανδία. Αλλά δεν είναι συζήτηση στην οποία συμμετέχει η Κομισιόν. Όπως είπατε, η Ολλανδική κυβέρνηση μία μέρα αποφάσισε κάποια όρια για να διακρίνει ε, το ποιος δικαιούται και ποιος δεν δικαιούται κοινωνική στέγη μετά από συζήτηση ετών, εάν θυμάμαι καλά, 7 ετών, το κατόφλι αυτό, μετά υπό κάποιους όρους, δηλώσαμε πως είναι συμβατό. Αυτό είπαμε, το κατόφλι αυτό είναι συμβατό. Υπό τους όρους της απόφασής μας του 2009, πριν ε, δηλαδή αναλάβω εγώ πώς μπορεί να παρέμβει η Κομισιόν στην ε, πολιτική της κοινωνικής στέγασης της Ολλανδίας. Μόνο εάν οι Ολλανδικές αρχές αλλάξουν το υπάρχον πλαίσιο, δηλαδή πρέπει να ε, ειδοποιήσουν πρώτα απ' όλα, να τα κοινοποιήσουν αυτά στην Κομισιόν γιατί Βεβαίως το πλαίσιο αυτό το είχαμε εγκρίνει με την απόφασή μα του 2009. Οπότε αν αλλάξει κάτι θα πρέπει να μας ειδοποιήσουν και τότε θα δούμε. Αυτό, αυτό είναι όλο. Ε, εντάξει, επαναλαμβάνω τα προφανή, τα προφανή για εσάς. Το είπα αυτό και σε κάποιου ε, ευρωβουλευτέ από διάφορε πολιτικές οικογένειες. Τους είπα ακριβώ τα ίδια πράγματα. Και τα ίδια ακριβώ και στην κυβέρνηση πρόσφατα ήρθαν σε επαφή μαζί μου και τους εξήγησα. Ο Γενικά μου διευθυντής ε, δεν είναι πολιτικός, είναι Ολλανδός, ήταν εδώ πέρα στο κοινοβούλιο, είπε ακριβώς τα ίδια. Ε, τα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα την πολιτική της Ολλανδίας. Όσον αφορά τις καταγγελίες, εάν δεν κάνω λάθος, το ζήτημα αυτό της απόφασης του 2009 εκρεμεί ενώπιον του δικαστηρίου και τα εμπλεκόμενα μέρη είναι και από τις δύο μεριές. Αυτοί που θεωρούν πολύ χαμηλό το κατόφλι και αυτούς το θεωρούν ε, πολύ ψηλό. Και οι δύο πλευρές νομίζω προσωπούνται στη διαδικασία. Μάλιστα. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο προς τις ε, δαπάνες των κυβερνήσεων. Στην Ευρώπη πάνω από το 50% του ΑΕΠ προέρχεται από το κράτος, ενώ στην ε, Κίνα είναι πολύ χαμηλότερο. Ποιος είναι ο καπιταλιστής και ποιος ο κομμουνιστής. Οι επόμενες δύο ερωτήσεις τώρα. Κυρία Πρόεδρε, σχετικά με τον κομμουνισμό, να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τον φόρο ε, οικονομικών συναλλαγών. Το θέμα αυτό συζητείται στην Ένωση, αλλά δεν φαίνεται να υιοθετείται. Από την άλλη, Δαρία και η Γερμανία ανέφεραν ότι είναι έτοιμες να το εισαγάγουν στην Ευρωζώνη, δημιουργώντας μια Ευρωπαϊκή Ένωση δύο ταχυτήτων. Αν λοιπόν εισαχθεί αυτός ο φόρος εντός της Ευρωζώνης και όχι εκτός, η ερώτησή μου αφορά τον ανταγωνισμό τι θα γίνει σε σχέση με το πεδίο. Τι θα γίνει δηλαδή ε, με τις επιχειρήσεις ε, εκείνες οι οποίες θα φύγουν από την Ευρωζώνη και θα πάνε εκτός Ευρωζώνης ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Συγκαπούρη ας πούμε. Αυτό θα είναι τεράστια απειλή για την Ευρωζώνη. Για σας, τον Επίτροπο Ανταγωνισμού, αυτός ο φόρος ε, οικονομικών συναλλαγών είναι συμβατός με τις αρχές τις οποίες πιστεύετε και θέλετε να προστατεύσετε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, κύριε Επίτροπε, να σας ευχαριστήσω για την εισήγησή σας. Μιλήσατε για ανταγωνισμό σε περίοδο κρίσης. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να υποβάλω την εξή ερώτηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή οι ιδιώτες να αποζημιωθούν για θέματα που άπτονται αυτού του τομέα. Είπατε ότι ίσως αλλάξει αυτή η κατάσταση, αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Πώς θα αλλάξει η κατάσταση αυτή και πώς συνάδει με την κατάσταση των επιχειρήσεων, διότι η Επιτροπή πολλές φορές επιβάλλει χρηματικές ποινές δεν είναι μεγάλος ο φόρτος για τις επιχειρήσεις. Επίσης, ως προς τους οίκους αξιολόγησης, στην πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή μιλάτε για αύξηση του ανταγωνισμού και μιλάτε για δυνατότητα σύγκρισης αξιολογήσεων ή ένα νέο βαθμολόγιο για τους οίκους αξιολόγησης. Νομίζετε ότι αυτό θα βοηθήσει την αγορά με όλες τις δυσκολίες που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και δεν, θεωρείτε ότι χρειάζονται άλλα μέτρα για να υπάρξει το άνοιγμα της αγοράς σε άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς. Ευχαριστώ. Σχετικά τώρα με το φόρο οικονομικών συναλλαγών, αυτή είναι μια πρόταση που εστάλει από την Κομισιόν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως ως μέλος του Κολεγίου των Επιτρόπων υιοθετώ απολύτως την πρότασή μας και υποστηρίζω πλήρως την πρόταση αυτή, αυτό το οποίο λέει δηλαδή η πρότασή μας. Αυτή είναι η θέση μου όχι μόνο υπό την ιδιότητά μου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο σύνολό της θα πρέπει να υιοθετήσει και να εισαγάγει αυτό το φόρο οικονομικών συναλλαγών. Τώρα, μια γενική θέση. Κρατικές ενισχύσεις, τρευλώσεις ανταγωνισμού και φορολογία. Σύμφωνα με το δόγμα, αλλά και την ομολογία, υπάρχουν στρεβλώσεις ανταγωνισμού όταν διάφορα επίπεδα φορολογίας υφίστανται εντός μιας χώρας μέλους και επιβάλλουν διακρίσεις ε, ε, ε, έναντι κάποιων οικονομικών φορέων μάλλον σε κάποιους οικονομικούς φορείς έναντι κάποιων άλλων. Αυτή λοιπόν η επιλεκτικότητα όταν ισχύει εμείς αντιδρούμε. Εάν όμως διαφορετικές χώρες μέλη έχουν διαφορετικά επίπεδα φορολογίας, θα έλεγα ότι βεβαίως θα θέλαμε ή θα, θα επιθυμούσαμε να αντιδράσουμε, αλλά δεν μπορούμε. Γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα φορολογίας που σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούν στρεβλώσεις. Διαφορετικά επίπεδα φορολογίας, ας πούμε, στην εταιρική φορολογία, στη φορολογία των εταιριών. Αλλά αυτές οι διαφορές όταν είναι μεταξύ χωρών μελών και όχι εντός μιας χώρας μέλους, εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε νομικά. Σχετικά με τη δική σας ερώτηση τώρα. Η επιβολή, η ιδιωτική επιβολή ανταγωνισμού και η κρατική επιβολή ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά. Απαιτείται όμως καλύτερο συντονισμός. Συντονισμός μεταξύ του ιδιωτικού και του κρατικού. Και ακριβώς αυτό το νόημα έχει η νομοθετική πρωτοβουλία την οποία ανακοίνωσα για το επόμενο, για το προσεχές έτος. Κατά τη γνώμη μου, η δημόσια παρέμβαση θα πρέπει να προηγηθεί. Δεν, δεν μπορώ να το επιβάλλω βέβαια αυτό, αλλά είναι καλύτερο. Ε, ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να λάβει υπόψη τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει το δημόσιο σκέλος, το κράτος δηλαδή. Αλλά εάν οι απαιτήσει οι απαιτήσει για αποζημίωση ή ε, αντιστάθμιση προλαμβάνει αυτές, αυτή την, ε, την απόφαση από τον κρατικό φορέα, εγώ ποτέ δεν θα θεωρήσω τις αντισταθμίσεις που τις αντισταθμίσεις που καταβάλλονται από τον ιδιωτικό φορέα ως παραβίαση. Δηλαδή, η αντιστάθμιση ή η αποζημίωση θα πρέπει να βασίζεται και να εδράζεται στην απόφαση ε, του κρατικού φορέα. Δηλαδή, στόχος μας δεν είναι να αποζημιώσουμε, στόχος μας είναι να τιμωρήσουμε αυτόν που παραβιάζει και να λειτουργήσουμε αποτρεπτικά ώστε να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Τώρα, σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς. Στην πολιτική ανταγωνισμού, οι πιο σημαντικές αποφάσεις είναι οι ατομικές αποφάσεις, οι, οποία, οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη. Σε κάθε απόφαση που υιοθετούμε έναντι των καρτέλς, έναντι της δεσπόζουσες θέσεις, Η επιβάλλοντας θεμελιώδεις αρχές της συγχωνεύσης παραδείγματος χάρη. Αυτές είναι ενέργειες που έχουν ως στόχο να αρθούν οι περιορισμοί, να αρθούν τα εμπόδια στην αγορά. Δηλαδή η πολιτική ανταγωνισμού θέλει να ανοίξει τις πύλες για νέες εισόδους αυτός είναι ο στόχος. Άρα λοιπόν η επιβολή κανόνων ανταγωνισμού βοηθά το άνοιγμα των αγορών και την κατάργηση των εμποδίων. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Επειδή αναφερθήκατε στο εταιρικό φόρο και τις διαστρεβλώσεις που μπορεί να υπάρξουν, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η βάση της φορολογίας είναι εξίσου σημαντική, διότι ε, είναι εύκολο να δει κανεί το ύψο τη φορολογία, αλλά είναι δύσκολο να συγκρίνει την αρχική βάση. Απάντηση. Συμφωνώ απολύτω, κυρία Πρόεδρε. Γι' αυτό ακριβώς και κάναμε τις προτάσεις που κάναμε και ελπίζω ότι εσείς και το Συμβούλιο ε, θα τα υιοθετήσετε αυτά που προτείνουμε το ταχύτερο δυνατό. Ωραία, αυτό θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Ο επόμενος συνάδελφος, παρακαλώ. Ο θα μιλήσω γαλλικά. Δύο ερωτήσεις. Έγινε μία έρευνα από την Κομισιόν για δόλιο χειρισμό του Euribor. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η έρευνα και του Libor. Δεν θα ήθελα να μπείτε σε λεπτομέρειες ως προς τις υποψίες σας, θα ήθελα όμως να δούμε περί τίνος πρόκειται, δηλαδή να δούμε τα γεγονότα και όχι τα ονόματα. Έχετε παρόμοιες έρευνες, διενεργούνται παρόμοιες έρευνες στο χρηματοοικονομικό σύστημα το οποίο υφίσταται συνέπειες, διότι αυτή η χειραγώγηση των επιτοκίων είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Το ΔΕΚ όχι εσείς δηλαδή, αλλά το ΔΕΚ δεν δέχτηκε έναν εταιρικό φόρο στο Γιβραλτάρ που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί αυτή η μεταρρύθμιση, η φορολογική μεταρρύθμιση σήμαινε παράνομη ενίσχυση των επιχειρήσεων. Εσείς το ερευνάτε αυτό, αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες για να δείτε κατά πόσο αυτά τα φορολογικά μέτρα υπέρ των επιχειρήσεων αποτελούν στρέβλωση στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Η Ελίσσα. Ευχαριστώ. Η πρώτη μου ερώτηση έχει έχει σχέση με αυτό που είπε ο Φιλίπ. Απογοητεύτηκα διότι στο πρόγραμμα για το 2012 δεν γίνεται λόγος για φορολογική, φορολογικό συντονισμό, τουλάχιστον για τις άμεσες φορολογήσεις, διότι αυτό στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Ως προς τις κρατικές ενισχύσεις τώρα, στον χρηματοοικονομικό τομέα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε, να διευθετήσουμε αυτές τις ενισχύσεις χωρίς να δούμε την τραπεζική κρίση. Γιατί οι τράπεζες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ταμείο για την επίλυση του ζητήματος, των ζητημάτων αυτών έτσι ώστε να γίνονται άμεσες κρατικές ε, παρεμβάσεις και αυτό αργεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σας πω τι ακολουθείτε, να σας ρωτήσω τι ακολουθείτε με τον Μπαρνιέ. Επίσης έχουμε τρεις οίκους που ε, δεσπόζουν στην αγορά, δηλαδή ελέγχουν το 96% της αγοράς και επειδή μιλάμε για τους ίδιους μετόχους δεν πρόκειται για στρέβλωση του ανταγωνισμού. Θα ήθελα να μου απαντήσετε και σε αυτό. Είναι ύψης της σημασίας ως προς τη συγχώνευση Euronext με τη Deutsche Börse και με το NYSE. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτό θα οδηγήσει σε διαφάνεια της αγοράς και θα χρηματοδοτηθεί πραγματική αγορά ή θεωρείτε ότι στρεβλώνει στοιχεία της αγοράς. Να απαντήσω ισπανικά ό,τι θέλετε, λέει η Ελίζα. Ευχαριστώ. Καταρχήν στα γαλλικά δεν μπορώ να σχολιάσω την πρώτη σας ερώτηση για το Euribor. Στο μέλλον, στο μέλλον τώρα δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Δεν μπορώ σήμερα. Ως προς την απόφαση του ΔΕΚ για το Γιβραλτάρ, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διότι παρακολουθήσαμε το θέμα και το δικαστήριο δέχτηκε την επιχειρηματολογία της Κομισιόν. Υπήρχε πράγματι διάκριση και επιλεκτική μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων στο Γιβραλτάρ και ήταν οι επιχειρήσεις offshore, υπεράκτιες δηλαδή. Δεν μιλάμε μόνο για διάκριση ως προς το επίπεδο φορολόγησης, το οποίο και αυτό αναγνωρίστηκε ως αντίθετο προς τους κανόνες ανταγωνισμού, αλλά είχαμε και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που μιλούσε για φορολογικούς παραδείσους που πρέπει να παταχθούν. Επειδή ακριβώς θα πρέπει να γίνει μια πιο ενδελεχής ανάλυση και εξέταση θεμάτων ε, διακρίσεων, φορολογικών διακρίσεων, υπό την ε, οπτική γωνία του ανταγωνισμού ζήτησα από τη Γενική μας Διεύθυνση να προετοιμάσει ένα έγγραφο για να συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δράση μας κατά των διακρίσεων αυτού του τύπου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις. Και επειδή ξέρω ότι ο κύριος Λαμπέρ παρακολουθεί αυτές τις συζητήσεις, θα τον ενημερώσω και εσάς και την Επιτροπή σας για τα συμπεράσματά μας. Και ελπίζω να μας υποστηρίξετε. Και απαντώντας στην κυρία Ιντβελτ, μιλάμε για περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης και το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο από πλευράς δαπανών αλλά και εσόδων, στον προϋπολογισμό δηλαδή. Ελπίζω να έχουμε πιο ενδελεχείς συζητήσεις κατά το 2012. Ελίσα. Ελίσα, τώρα, όταν μιλάμε για φορολογικό συντονισμό, ε, θα σου επαναλάβω αυτό που είπα και στον κύριο Λαμπέρ. Δεν μπορούμε να ορίσουμε τη φορολόγηση των κρατών μελών, ούτε μπορούμε να αποφανθούμε νομικά. Τη στιγμή που υπάρχει όμως μεγαλύτερος ο φορολογικός συντονισμός, τότε οι φορολογικές τρευλώσεις μειώνονται και ιδιαίτερα μέσω του συντονισμού που σημαίνει πολιτική θέληση όσων συντονίζουν, δηλαδή των κρατών. Μπορούμε να φτάσουμε λοιπόν σε αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούμε να επιτύχουμε μόνο μέσω των κρατικών ενισχύσεων. Διότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση από τις κρατικές ενισχύσεις. Κάθε χώρα έχει τη δική της αγορά, τη δική της δυναμική αγοράς. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν γίνονται στρεβλώσεις ιδιαίτερα με τις γείτονες χώρες και μπορούμε με το συντονισμό να άρουμε στρεβλώσεις. Το ΕΚΟΦΗΝ δημιούργησε την ομάδα Πριμαρόλο, όπως ονομάζεται, έτσι ώστε να άρουμε φορολογικά μέτρα τα οποία είναι επιζήμια. Εγώ δεν, έχω, δεν φέρω αυτή την ευθύνη αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να σας πω πώς έχουν οι συζητήσεις αυτής της ομάδας η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνει τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. Πώς να αντιμετωπίσουμε την κρίση των τραπεζών. Οι κρατικές ενισχύσεις είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση, όμως δεν είναι το μέσο που ε, μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως. Βεβαίως υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις, αλλά χρησιμοποιούμε αυτό το μέσον και για, γιατί δεν υπάρχουν μηχανισμοί πλήρους εξυγίανσης. Δεν θέλω να δώσω παραδείγματα. Όταν εγκρίνουμε μία ε, τραπεζική εξυγίανση, απαιτούμε επενδύσεις, αλλαγές στο business model και συγκεκριμένους όρους για την κατανομή των βαρών και ούτω καθεξής. Ένα μέρος αυτών των αποφάσεων αντιστοιχεί στους μηχανισμούς εξυγίασης που δεν υπάρχει. Ο Μισελ Μπαρνιέ σήμερα προετοιμάζει μία πρωτοβουλία, δηλαδή ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, μηχανισμούς ευρωπαϊκής εμβέλειας. Υπάρχουν σε ορισμένα κράτη-μέλη, δεν υπάρχουν όμως σε ευρωπαϊκή κλίμακα και τη στιγμή που έχουμε μία διασυνοριακή διαφορά υπάρχουν επιπρόσθετες διαφορές. Η Ελίζα, ακόμα και σε περίπτωση ανταγωνισμού θα πρέπει να δούμε και τις χώρες που ελέγχει η Τρόικα. Υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού διότι το τραπεζικό σύστημα αυτών των κρατών είναι διαφορετικό. Οι χώρες αυτές, τις οποίες ελέγχει η Τρόικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δουνουτού, εδώ υπάρχει ειδική εποπτεία για να δούμε κατά πόσο πληρούνται οι όροι κρατικών ενισχύσεων, αλλά μας ενδιαφέρουν οι γενικότεροι κανόνες. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τις ε, χώρες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες και εδώ είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί ως προς αυτές τις χώρες. Ως προς τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι γεγονός ότι επειδή έχουμε 30 εγγεγραμμένους οίκους στην ΕΣΜΑ, υπάρχουν όμως τρεις μεγάλοι οίκοι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αυτοί οι μεγάλοι Υπάρχουν δύο οίκοι που είναι μεγαλύτεροι από τον τρίτο. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα αντιτράστα. Δεν πρόκειται για ε, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Όταν αναλύσουμε την κατάσταση των οίκων αξιολόγησης φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται μια ρύθμιση, κάτι το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα. Για τρίτη φορά ορίσαμε αυτό το πλαίσιο των οίκων Εγώ, η γενική μου διεύθυνση, έχει αναλύσει όλες τις ε, πτυχές της ε, δυσλειτουργίας των οίκων αξιολόγησης και είναι πολλές αυτές οι πτυχές αλλά σε καμία περίπτωση δεν βρήκαμε λύσεις που προέρχονται από το αντιτράστ, από περιπτώσεις αντιτράστ. Γιατί σε αυτή την περίπτωση διενεργείται έρευνα και αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Θέλουμε δηλαδή να ικανοποιήσουμε την κατάσταση με βάση αυτή τη λειτουργία Εν πάση περιπτώσει, η λειτουργία των οίκων δεν είναι ικανοποιητική και πολλές φορές ε, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιλύουν. Αλλά στην πρόταση που εγκρίναμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θέλουμε να ανοίξουμε ένα, το άρθρο 102, μία έρευνα δυνάμει του άρθρου 102. Μας ενδιαφέρουν οι συγκρούσεις συμφερόντων ή πολλές φορές έλλειψη διαφάνειας στη μεθοδολογία ή έλλειψη διαφάνειας για να δούμε πώς ορίζουν τον κίνδυνο και πώς τον επιλύουν. Αλλά δεν είναι θέμα αντιτράστη. Είναι θέματα άλλου είδους που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Τέλος, ως προς τη συγχώνευση του New York Stock Exchange, του Euronext και της Deutsche Börse. Αυτό ε, ερευνάται τώρα και είχαμε συζητήσεις ήδη από το Φεβρουάριο για αυτή την ενδεχόμενη συγχώνευση. Την προηγούμενη Παρασκευή λάβαμε μία πρόταση αντιμετώπισης για να προσπαθήσουμε να άρουμε τις διαφορές που υπάρχουν. Πρόκειται για σοβαρές αντιρρήσεις από τη δική μας πλευρά και το ξέρουν τα εμπλεκόμενα μέρη. Αναλύουμε τα μέτρα που μας πρότειναν τα εμπλεκόμενα μέρη το, την Παρασκευή θα γίνει μία δοκιμασία της αγοράς και τη στιγμή που προβλέπονται ρυθμίσεις θα δούμε τι θα γίνει μεταξύ 22 Δεκεμβρίου και 23 Ιανουαρίου. Στις 23 Ιανουαρίου θα λάβουμε απόφαση με βάση τις αντιρρήσεις που προβάλλουμε. και θα δούμε τι θα γίνει υπό το φως των λύσεων ή των μέτρων που προβλέπουν τα εμπλεκόμενα μέρη. Could I tempt you instead of... Ε, αντί να δείτε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι γενικότερο για την ε, προτινόμενη υποδομή καθώς έχουμε το εμίρκετο και, τη μύφη την οδηγία ε, μπροστά μας και ποιο είναι το όραμά σας όσον αφορά την ε, πρόσβαση και τις προδιαγραφές γιατί προφανώς υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της νομοθεσίας ε, των χρηματοοικονομικών και κάποιων γενικών αρχών του ανταγωνισμού. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες γιατί η υπόθεση αυτή ακόμα εκκρεμεί και δεν μπορώ να αποκαλύψω λεπτομέρειες μπορώ να σας πω πως η σχέση μεταξύ η, μεταξύ της ε, προτινόμενης συγχώνευσης Nice ε, Euronext και Deutsche Börse και της νομοθεσίας που συζητιέται στο Συμβούλιο αφορά περισσότερο το MIFIR, το MIFID 2 παρά το EMIR ως νομοθεσία γιατί το EMIR έχει περιοριστεί σε παράγωγα over the counter και οι περισσότερες ε, αντιρρήσεις μας ε, πηγαίνουν ε, πιο πολύ όσον αφορά την εμπορία παραγωγών σε ένα χρηματιστήριο. Δεύτερον, χωρίς να αναφερθώ στην συγκεκριμένη περίπτωση, μπορώ να σας πω πως οι διατάξεις οι οποίες περιέχονται στο μυθιτίο και το Μύφιτ. συμφωνούν πλήρω με την άποψή μου του πώς πρέπει να λειτουργεί αυτή η αγορά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω πως είναι δύσκολη η θέση σας. Οι επόμενες δύο ερωτήσεις, ε, και ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ πως ε, πρέπει να σας ευχαριστήσω και εξ ονόματος και ο για το θέμα των συνταξιδοτικών όσον αφορά αυτά τα οποία αναφέρατε για το επιέλα και των κατοφλίων και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι για το πόσο μεγάλη διαθεσιμότητα δείχνεται καθώς δεν είσαι υποχρεωμένος, αλλά δείχνεται πάντα πάρα πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα και σας ευχαριστούμε. Ε, μία ερώτηση όσον αφορά την έκθεση και το πλαίσιο το οποίο συζητιέται εκεί πέρα για τις, υπηρεσίες, τις οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Μιλάμε για ένα πλαίσιο ποιότητα το οποίο θέλετε να θέσετε. Όχι το πλαίσιο που σου ζητάνε οι σοσιαλδημοκράτες και οι λοιποί σύμφωνα στο άρθρο 14, αλλά ένα ποιοτικό πλαίσιο. Μπορούμε να το περιμένουμε αυτό μέσα στο έτος ε, πώς ε, έχει το χρονοδιάγραμμα. Κατόπιν ένα άλλο ερώτημα σε σχέση με, το, με αυτό το οποίο είπε η κυρία Ενετφέλτ, στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω. Γιατί εγώ ακούω συνεχώς μία φήμη πως εξακολουθεί να υπάρχει η ίδια άποψη στους εμπλεκομένους. Όλοι λένε πως η Κομισιόν ανάγκασε την Ολλανδία να θέσει αυτά τα όρια και η Κομισιόν θέλει να καταστρέψει έτσι την κοινωνική στέγη. Η Κομισιόν ξεκίνησε στην Ολλανδία και θα τα συνεχίσει αυτά αλλού. Μετά τη συζήτησή μας βεβαίως βλέπω πως αυτό δεν συμβαίνει. Ήδη ε, το έχετε πει, αλλά θα ήθελα πραγματικά να ξεκαθαρίσετε πως το κατόφλι αυτό το όρισε η Ολλανδία και όχι η Κομισιόν. Αυτό θα μας βοηθούσε πάρα πολύ ε, για όλους τους ενδιαφερόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα τρίτο ερώτημα για τις υπηρεσίες, ε, της οίκους αξιολόγησης ο Ρόλαντ Μπέργκερ ερεύνησε την ιδιοκτησία των οίκων αυτών αξιολόγησης και χρειάστηκε αρκετές ομάδες για να καταλάβει τι ανήκει σε ποιον. Και το ενδιαφέρον είναι πως οι ιδιοκτήτες της ε, Standard Poor's δεν είναι πως ε, συνδέονται όλοι μεταξύ τους ε, και με την Moody's, αλλά υπάρχει και μεταξύ των δύο ομάδων μια σύνδεση και βλέπετε πως είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι υποφελούνται ε, πάρα πολύ όταν αλλάζει μια αξιολόγηση. Οπότε το θέμα της κατάξυσης της θέσης τους ε, ε, νομίζω πως εδώ πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Νίκλας. Κύριος Καλημέρα κύριε Αλμούνια αν έχετε δέσει γερά τη ζώνη ασφαλείας σας, ας πάμε από την Ολλανδία λίγο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν συζητείται έντονα το θέμα των ειδικών οικονομικών ζωνών. Κατά την τελευταία επίσκεψη του Αντικαγκελαρίου της Γερμανίας αλλά και του Υφυπουργού Οικονομικών εξετέθη, προβλήθηκε αυτή η ιδέα και αναφέρθηκε ότι συνεξετάζεται με την Κομισιόν. Δηλαδή ειδικέ οικονομικές ζώνες, η ιδέα της Γερμανίας συνεξετάζεται μαζί σας, με την Κομισιόν. Σας ερωτώ λοιπόν, πράγματι ασχολείστε με αυτό το θέμα. Συζητάει δηλαδή η Κομισιόν την ίδρυση ειδικών οικονομικών ζωνών ή την αλλαγή του νόμου περί επενδύσεων στην Ελλάδα. Συζητάτε ειδικά κίνητρα φορολογικά, εργασιακά, ποια θα είναι αυτά. Και αν έτσι έχουν τα πράγματα, όλο αυτό είναι συμβατό με τα κοινωτική συγγνώμη, νομοθεσία και τα περί ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Eh. Ευχαριστώ. Στον κύριο Σάιμον επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχική μου εισήγηση. Ε, εκτίμησα ιδιαίτερα την έκθεσή του. Απομένουν λίγες εβδομάδες πριν λάβουμε την τελική απόφαση για το νέο πακέτο οικονομικών υπηρεσιών γενικού ε, ενδιαφέροντος και σε αυτή την έκθεση ένα από τα θέματα είναι οι κανόνες de δηλαδή τα κατόφλια που ορίζουμε κάτω από τα οποία δεν υπάρχει ε, ενίσχυση και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες ε, δεν έχουν υποχρέωση έγκαιρης προειδοποίησης πριν από την χορήγηση ενισχύσεων. Χρησιμοποιούμε, βλέπουμε την επιχειρηματολογία και θα λάβουμε μια απόφαση. Αλλά θα ήθελα να πω ότι η έκθεση ε, συμπίπτει ως προς την, ε, τις απόψεις. Θα λάβουμε υπόψη λοιπόν αυτά τα κατόφλια σοβαρά και όλα τα στοιχεία που μας ε, βοηθούν για την, τον ορισμό των κατοφλίων. Ως προς το θέμα της ποιότητας, αυτό έχει σχέση με άλλη πρωτοβουλία της Κομισιόν που δεν είναι δικής μου ε, η υπευθυνότητα. Θα σας τα αναλύσει ο Μισελ Μπαρνιέ το απόγευμα. Η κυρία Ιντβέλτ δεν είναι εδώ. Μπορείτε να της πείτε ότι της απαντώ το ίδιο. Το ίδιο που είπα και για την Ολλανδική κυβέρνηση και όπως είπα και σε άλλες ομάδες και κράτη. Ως προς τα κατόφλια για θέμα κοινωνικής στέγης, τα κατόφλια αυτά τα ορίζουν οι Ολλανδικές αρχές και μόνον. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να αναλύσει κατά πόσο αυτά που αποφάσισαν οι Ολλανδικές αρχές είναι συμβατά ή όχι με το κοινοτικό δίκαιο ποτέ δεν θα υπάρξω Ολλανδός πολιτικός. Ως προς τους οίκους αξιολόγησης, ούτε, ούτε, ούτε Γερμανός, ούτε Γερμανός πολίτης. Αυτό θα ήταν το δεύτερο αίτημά μου. Μετά τη δική μου υπηκότητα θέλετε, αλλά την γερμανική. Ως προς τους οίκους, επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην κυρία Φερέιρα. Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν μεγάλα προβλήματα. Και ένα από τα μεγαλύτερα αντιμετωπίζεται με την πρόταση της Κομισιόν και θα το συζητήσετε το Συμβούλιο. Μιλάμε για σύγκρουση συμφερόντων εδώ είναι ένα θέμα που ενυπάρχει και το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί κάπως. Δηλαδή θα πρέπει να απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Εάν εσείς πρέπει να ορίσετε κάτι, δεν μπορείτε να είσαστε πελάτης αυτού του οργανισμού. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα άρθρα 101 και 102 των συνθήκων. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα δύο άρθρα. Τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να ορίσουμε τους κανόνες ανταγωνισμού με βάση τα άρθρα 101 και 102 είναι πολύ σημαντικά. Δεν το αρνούμε αυτό, διότι εγώ πρέπει να εφαρμόσω αυτά τα δύο άρθρα μίλησα λίγο πριν για τη συγχώνευση της Deutsche Börse με τη Euronext και την ε, NYSE. Μιλάμε για συγχώνευση 9 δις. πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανόνες ε, του ανταγωνισμού. Όταν έχουμε ένα τέτοιο μέσο, δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε για οποιαδήποτε στόχο. Θα πρέπει να εφαρμοστεί εκεί που πρέπει. Διαφορετικά αποδυναμώνουμε το μέσον αυτό, το μηχανισμό αυτό και δεν φτάνουμε στο στόχο μας. Το πρόβλημα των οίκων αξιολόγησης δεν αφορά θέματα αντιτράστ. Το, το τονίζω αυτό. Υπάρχουν θέματα σύγκρουση συμφερόντων, όχι θέματα αντιτράστ. Και, και το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά. Λίγες μέρες πριν έγινε λόγος για καρτέλ η εικοναξιολόγηση, μα δεν είναι καρτέλ. Όσο άσχημα και να τα πηγαίνουν και με τα σφάλματα που έχουν διαπράξει, δημιουργούν και μεγάλη ζημία, ζημιώνουν την αγορά. Και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά. Αλλά δεν πρόκειται για παραβίαση των άνθρων 101 και 102. Τη στιγμή πως υπεύθυνο θεμάτων ανταγωνισμού δω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για την εφαρμογή των άρθρων αυτών, 101 και 102, θα δράσω άμεσα, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το μέσο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρύθμιση, μια διαδικασία ρύθμισης, όπως προτείνει η Επιτροπή. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όμως τα άρθρα 101 και 102. Για τον κύριο Χουντή τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα σε σχέση με αυτές τις δύο ζώνες. Η μόνη διαφορά μεταξύ ζωνών αφορά, ορίζεται από τα 17 κράτη που έχουν ένα νόμισμα, το ευρώ, και πρόκειται για τα κράτη που ορίζουν αυτό τον τρόπο λειτουργίας. Εμείς ως Κομισιόν συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση της τελευταίας δόσης και ο κύριος Παπαδήμος, όπως ξέρετε, μίλησε με τους Μπαρόζο και Βαν Ρομπόη και ελπίζω τα πράγματα να επιληθούν το ταχύτερο δυνατόν, ειλικρινά το εύχομαι, εμείς έχουμε ορίσει μια task force για να χρησιμοποιήσει κατά το μέγιστον τα μέσα που διαθέτουμε ως Ευρωπαϊκές Αρχές για να ευεργετηθεί η Ελλάδα, ελπίζω με θετικά αποτελέσματα και δεν πρέπει να υπάρχουν οικοτολογίες, γιατί αυτό δεν βοηθάει κανέναν και δεν υπάρχει καμία, δεν είναι βάσιμες αυτές οι κοτολογίες. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Ακόμα μια ερώτηση που θα ήθελα να θέσω στον κύριο Επίτροπο. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχουν επιτόκια κάτω, πάνω από 4% σε αυτή την ε, περίοδο κυβερνητικής αλλαγής. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχει στρέβλωση της, ε, ε, του ελεύθερου ανταγωνισμού. Εγώ διάβασα τις απαντήσεις σας στις γραπτές μας ερωτήσεις και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να επαναλάβω αυτές τις γραπτές ερωτήσεις. Έχω όμως την εντύπωση ότι είμαστε αδύναμοι γιατί μιλάμε και για το ρόλο των ε, οίκων και μου λένε εσύ τι κάνεις ως Ευρωβουλευτής με τις ε, γραπτές ή προφορικές σου ερωτήσεις. Δεν θα μπορούσε η Κομισιόν να δράσει πιο αποφασιστικά έτσι ώστε αυτές οι κάκιστες πρακτικές να μην επαναληφθούν. Απάντηση. Δεν έχω εδώ όλες τις ε, γραπτές απαντήσεις σας που μου απαστήλατε για αυτές τις ερωτήσεις και το μόνο που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Ε, αν γνωρίζω καλά, στην Ισπανία υπάρχει μία ρύθμιση για τα όρια των πολιτικών στοιχείων παθητικού που μπορούν να οριστούν, οριστούν με τη δημόσια βοήθεια ή αρρωγή. Γιατί στην προεκλογική περίοδο και μετά θα πρέπει να τηρείται το γράμμα του νόμου. Και αυτό αφορά και τον τραπεζικό τομέα. Τη στιγμή όμως που υπάρχουν διαφορές και χτες μιλήσαμε και για την Banco και εμείς δώσαμε μία προσωρινή αδειοδότηση. Στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ισπανίας ή άλλου κράτους μέλους, μέσα στα πλαίσια έξι μηνών, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να απαντήσει στην Επιτροπή με βάση ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης. Και στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ισπανίας και της Ευρώπης, δηλαδή στη περίπτωση που αναφέρεται θα υπάρξει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης και ένα από τα στοιχεία τα οποία αναλύονται και που μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι η πολιτική αναδιάρθρωση στοιχείων παθητικού. Και εδώ πολλές φορές έχουμε επιβάλει περιορισμούς τη στιγμή που το σχέδιο αναδιάρθρωσης συζητείται και εγκρίνεται εδώ. Μέχρι τώρα στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ισπανίας που λάβαν χρήματα. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που να έχει ε, αποφασιστεί. Γιατί στην περίπτωση της Καστίγια Λαμάντσα δεν έχει ληφθεί απόφαση και για τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή δεν έχουν παρέλθει έξι μήνες ή οι ενισχύσεις τύπου FROB 1 έλαβαν χώρα σε επίπεδο μείον 2% και αναλύσαμε την βιωσιμότητα του σχεδίου που υποβλήθηκε. Από την 1η του 2011 οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση θα υπόκειται σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης. Και όταν μιλάμε για σχέδια αναδιάρθρωσης συγκεκριμένα, θα μπορείτε να υποβάλλετε περισσότερες ε, ερωτήσεις και θα σας απαντήσω αναπερίπτωση. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ πέρα τελειώνει η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Επίτροπο. Δεν είμαι σίγουρος εάν ε, μας υποσχεθήκατε ότι θα ξανάρθετε, αλλά συνήθως είστε ετοιμόλογος. Σας ευχαριστώ πολύ και βεβαίως αναμένω να σας ξαναδούμε του χρόνου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. εχουμε Έχουμε ε, ένα-δυο λεπτά για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην παρουσία. Θα περιμένω για να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Ωραία, σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης που πρόκειται για την ε, οδηγία 2003-71 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών δίνω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στις 11 Οκτωβρίου θεώρησα σημαντικό να κάνουμε μια δεύτερη συζήτηση για το θέμα αυτό, καθώς η ψηφοφορία πριν από τα Χριστούγεννα ούτως ή άλλως αναβλήθηκε και αυτό έγινε, θέλω να τονίσω, σε συμφωνία με τις υπόλοιπες ε, πολιτικές ομάδες, ε, καθώς είχαμε βεβαίως την οδηγία περιφερειακότητας 2, ε, 400 εκείνες σελίδες που μας έστειλε αρχές Νοεμβρίου η Κομισιόν. Ήταν οπωσδήποτε θετικό το ότι αναμείναμε τις εφαρμοστικές ε, διατάξεις για να έχουμε μια συνολική άποψη της ε, Γενικής ε, Οδηγίας. Οπότε για λόγους και τυπικούς και ουσιαστικούς είναι λογική η κίνηση αυτή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σκεφτούμε σε ποιο βαθμό τα πλαίσια αυτά θα πρέπει να ε, συμφωνούν με την οδηγία πλαίσια. Εδώ πέρα η Κομισιόν μιλάει για συνολικό πακέτο, αλλά πριν γίνει αυτό θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι τα κομμάτια που περιέχονται σε αυτό το πακέτο. Στις 9 Νοεμβρίου η Κομισιόν απέστειλε μια τεχνική ενημέρωση για τις εφαρμοστικές διατάξεις. Έγινε μια ενημέρωση στην οποία ήταν προσκεκλημένοι όλοι οι βουλευτές της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Ήταν μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση και θεωρώ πως είχε μια πολύ καλή συζήτηση. Η πρόταση των εφαρμοστικών διατάξεων και οι εξηγήσει της ε, Κομισιόν οπωσδήποτε θα μας βοηθούσουν για να βρούμε έναν ε, συμβασμό. Και εδώ πέρα βεβαίως εννοώ το θέμα των μακροπρόθεσμων εγγυήσεων. Έχουμε λοιπόν τα διάφορα ασφάλιστρα τα οποία είναι αυτό το αντικυκλικό και της ρευστότητα, ειδικά αυτό της ρευστότητα νομίζω είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να μην μεταβάλω απόψη, αλλά λαμβάνω υπόψη πως η πλειοψηφία των συναδέλφων οι οποίοι ε, έλαβαν το λόγο ήταν υπέρ ενός αντικυκλικού ασφαλίστρου. Θα πρέπει όμως να είναι σαφές πως με ένα τέτοιο ασφαλίστρο πλέον ε, υπάρχει και ο κίνδυνος ε, των credit spread risks. Όσον αφορά δε το ασφάλιστρο το λεγόμενο matching ε, premium ε, εξακολουθώ να είμαι επιφυλακτικός καθώς ε, θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μια διασφάλιση υπομορφή ενεργητικών στοιχείων της εταιρεία και αναρωτιέμαι πραγματικά εάν εδώ πέρα πράττουμε ορθά όταν ακριβώς υπονομεύουμε την συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών. Με τις δε τροπολογίες δεν είναι σαφές ε, ποια είναι η άποψη της πλειοψηφίας της Επιτροπής. Ο κατάλογος μέτρων της ε, Κομισιόν ε, για να περιοριστεί η τεχνητή ε, κινητικότητα οδηγεί νομίζω σε ένα συμμετρικό μηχανισμό προσαρμογής όσον αφορά τους ε, κινδύνους των μετοχών. Οπότε το ζήτημα είναι πώς ε, διασφαλίζουμε πώς τα μονομένα αυτά κομμάτια θα είναι συνεκτικά μεταξύ τους. Αυτά, κατά την άποψή μου, είναι τα ουσιαστικά ζητήματα, ειδικά δεδομένου του ότι ειδικά το ασφάλιστρο της ε, ρευστότητας θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εξέτασης. Επίσης αναφέρθηκε το ζήτημα των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε με τα κρατικά ομόλογα, τα οποία βεβαίω μα απασχολήσαν στην Επιτροπή μα. Από την πλευρά τη ε, Κομισιόν είχαμε ένα θετικό μήνυμα για μια λύση για ολόκληρο τον ε, κλάδο. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι σημαντικό ειδικά εδώ να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση και θα ήθελα να προσθέσω πως ε, κατά την άποψή μου θα άξιζε τον ε, λόγο, τον κόπο να προδιαγράψουμε τις εξελίξεις ειδικά στον τομέα των ε, ασφαλιών ε, και ειδικά να επέμβουμε στον ίδιο χρόνο μαζί με τις τράπεζες όσον αφορά τις απαιτήσει της κεφαλαϊκές. Εδώ πέρα βέβαια θα θέλαμε να τοποθετηθεί ξανά η Κομισιόν. Θεωρώ πως αυτά είναι τα βασικότερα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στην έκθεσή μας. Τα ανέφερα, αναμένω την άποψη των συναδέλφων και πραγματικά αναμένω την αξιολόγησή σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. And also... Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνεδρίαση που είχαμε ε, σχετικά με την εφαρμογή, διότι πράγματι είναι από απόϊχος αυτών που κάναμε εδώ. Και τώρα δίνω το λόγο στους Κιώδης. Καταρχήν ο Πίτερ. Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ τον Μπέρκ για τη σκληρή δουλειά. Και συμφωνώ μαζί σας, Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομιζιό, διότι έφερε τα μέτρα έγκαιρα και είναι πολύ χρήσιμο να κάνουμε μία εξέταση παράλληλη και αυτό με βοηθά να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα και να τα περιλάβω σε τροπολογίες. Πρώτον, υπέβαλα τροπολογίες μετά από διαβούλευση με πολλούς ε, εμπλεκόμενους κλπ. Για, για να δούμε αν το έγγραφο του επίπεδου 1 θα επηρεαστεί και σε ποιο βαθμό. Νομίζω ότι ο Κάρντ έχει λάβει υπόψη τις ε, τροπολογίες μου και έχει αντιληφθεί το νόημά τους. Καταρχήν, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ρήτρα ε, ασφαλείας ε, που και όταν κανείς συναντά ανθρώπους στην ΑΙΟΠΑ πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι αυτή είναι μια εξέταση εντός του Κοινοβουλίου και ε, δεν ε, λύνουμε τα πάντα ε, εν μια ανοιχτή. Είναι τεχνικά θέματα, ας πούμε ρυθμίσεις σε τεχνικό επίπεδο και αναζητούμε την πιο πρακτική προσέγγιση. Φανταστείτε να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση το 2009, την εποχή ε, που εξετάζαμε την Λισαβόνα. Δεν πρόκειται για καμία ε, καμία συνωμοσία και κανένα, μάλλον κανένα σχέδιο συνωμοσία. Απλώς πρέπει να λάβουμε υπόψη τις νέες συνθήκες. Η νέα προσέγγιση η οποία ε, προτείνεται είναι σημαντική και το Κοινοβούλιο θα έχει το ρόλο του. Λοιπόν, Είμαι της άποψης ότι ο συνδυασμός των ασφαλίστρων είναι πολύ σημαντικό για να εφαρμοστούν τα μέτρα. Υπάρχει μια σειρά κυκλικών προτάσεων που ασφαλώς θα ληφθούν υπόψη για το έγγραφο σε επίπεδο 1. Εάν θέλουμε δηλαδή να λάβουμε υπόψη αυτή την κυκλικότητα και αν είμαστε υπέρ της κυκλικότητας. Εμείς λοιπόν ως Κοινοβούλιο πιέζουμε καταρχήν και εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει όχι μόνο ο κλάδος, αλλά και οι τελικοί χρήστες αυτών των προϊόντων. Δηλαδή οι άνθρωποι θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερα ασφάλιστρα, αν δεν τα κάνουμε σωστά. Δεν είναι θέμα ελαστικότητας. Το έχουμε και ασφάλιστα αντικυκλικότητας. Και αυτά όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και την μακροοικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει δηλαδή να έχουμε μια ισόρροπη προσέγγιση, αντί να πούμε ότι το ένα πράγμα αφορά τη μία χώρα, το άλλο την άλλη και δεν μας ενδιαφέρει. Όχι όταν συναντάει κανείς εκπροσώπους του κλάδου ε, μας λένε ότι έχουμε μία, πέντε εργαλεία στη διάθεσή μας για να εφαρμόσουμε ε, αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Και αυτά δεν αρκούν. Αφήστε μας λοιπόν να προχωρήσουμε όπως εμείς γνωρίζουμε. Και επίσης δεν θα πρέπει να σκοτώσουμε, να εξαλείψουμε δηλαδή τις συντάξεις με αυτά τα οποία θα κάνουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. και επίσης είμαι έτοιμος να ε, υιοθετήσω και κάποιες θέσεις της εισηγήτριας, διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάτι που η Κομισιόν και η ΑΙΟΠΑ θα βασίζονται σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Και τέλος, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι διέγραψε το θέμα της, των προδιαγραφών, προδιαγραφών ισχύω τρίτης χώρας, διότι η εφαρμογή μέτρων με βάση τις προδιαγραφές δεν αρκεί. Δεν τα είχαμε πριν δεν τα είχαμε δει και διαρωτώ για ποιο λόγο έπρεπε να μπουν σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό θα ήθελα και να ζητήσω κάποιες εξηγήσεις από αυτού. Η Σιλβή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Μπουρκάρτ για το έργο που συνεχίζεται και ευχαριστώ και την Κομισιόν διότι το έγγραφο που εξέδωσε μας βοηθά. Εντάξει, είναι μακρύ, είναι σύνθετο, ε, θα προσπαθήσουμε να κολυμπήσουμε μέσα σε όλα τα τεχνικά, αλλά πάντως ελήφθησαν υπόψη κάποια από τα αιτήματά μας και ευχαριστούμε. Δύο σχόλια. Πρώτον, το, η κρίση επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες και ε, λαμβάνουμε μέτρα τα οποία είναι ενδεχομένως τεχνικής φύσεως αλλά θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες σε τομείς και στην αποταμίευση μακροπρόθεσμα. Στη Γερμανία πριν από μερικές μέρες συζητούσαμε έναν επενδυτή που έλεγε ότι όταν ε, κοιτά κανείς ποια είναι, ποιοι είναι οι μηχανισμοί που έχει στα χέρια του ένας επενδυτής θα δει ότι είναι ήδη σχέσεις που δεν είναι αξιόπιστες ή είναι ε, κρατικά ομόλογα τα οποία όμως δεν αποδίδουν επαρκώς και γενικότερα η αγορά είναι τόσο διαταραγμένη που οι επιπτώσεις ε, επί της πραγματικής οικονομίας επιδεινώνονται. Γι' αυτό λοιπόν λέω και επαναλαμβάνω ότι Χρειάζεται ισορροπία όχι μόνο μεταξύ των εμπλεκομένων, αλλά επίσης και μια, απαιτείται μια προσπάθεια για να διατηρήσουμε έστω μεσοπρόθεσμα αλλά και μακρυπρόθεσμα αυτά τα οποία έχουν αποκτηθεί με μεγάλη δυσκολία. Τώρα, σχετικά με την επιλογή των διαφόρων ε, μηχανισμών που έχουμε στη διάθεσή μας και την επιλογή ασφαλίστρων ε, ρευστότητας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην επιτρέψουμε ας πούμε ε, τοπικούς ή εθνικούς, ε, εθνικές ρυθμιστικές αρχές να παρέμβουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα, υπενθυμίζοντας όλα όσα είπε ο προλαλής σας. Βέβαια οι καταστάσεις είναι πολύ διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Θα πρέπει όμως να είμαστε βέβαιοι ότι το σύστημα θα παραμείνει επαρκώς διάφανο ούτως ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστές να μπορούν να λειτουργήσουν σε λίγο πολύ ισοδύναμο ή ισότιμο περιβάλλον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Μπέκαρτ ε, για τη σκληρή δουλειά που κατέβαλε ε, για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα. Ε, θα αναφερθώ στην ομιμότητα του περιεχομένου της παραγράφου 138 η ΑΙΟΠΑ είναι ένας φορέας ευρωπαϊκός. Δεν έχει όμως την αρμοδιότητα να λάβει αποφάσεις για, γενικές, για αποφάσεις γενικής εφαρμογής. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Έχω δώσει στον Μπέρκαρτ κάποιες εναλλακτικέ. Ας πούμε, κατευθυντήριες γραμμές για το πώς οι εθνικοί επόπτες θα λαμβάνουν αποφάσεις σε έκτακτες περιπτώσεις. Αυτή θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη κριτηρίων, αλλά ε, και νομίζω ότι αυτό θα, βοηθήσει τους εθνικούς επόπτες. Ένα άλλο θέμα είναι τα αντικειμενικά κριτήρια, το πότε η ΑΙΟΠΑ θα ε, θεωρεί ότι κάτι είναι έκτακτο και εξαιρετικό. Τώρα, σχετικά με τα κατώτατα όρια ή τα κατόφλια, δεν νομίζω ότι βοηθούν. Κατά την άποψή μου, οποιοδήποτε τιμή αναφέρεται θα πρέπει να εδράζεται σε μια ε, προηγούμενη αξιολόγηση. Η εποπτεύουσα αρχή θα πρέπει να αποφαίνεται κατά τακτά διαστήματα, ας πούμε ένα τρίμηνο ή Επίσης, η περίοδος εφαρμογής της ρήτρα θα, πρέπει να ε, διαρκεί τουλάχιστον τρία χρόνια και βεβαίως Μπέρχαρ ξέρω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά δυσχερές ε, θέμα, ε, φάκελο και γι' αυτό έχει την απόλυτη στήριξή μου. Ευχαριστώ. θα μιλήσω γερμανικά. Ευχαριστώ και εγώ τον Μπουρκχαρτ. Δουλε... Δούλεψε πάρα πολύ εδώ πέρα αλλά ξέρετε πως ε, αυτά τα οποία μας αυτά τα οποία αφορούν τα συναισθηματικά μπορούμε να τα πούμε στα γερμανικά. Οπότε τώρα θα μιλήσω αγγλικά. Πρώτον, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε τα εφαρμοστικά μέτρα και πράγματι είναι ενδιαφέρον ανάγνωσμα ε, του σχέδιου έκθεσης και μπορώ να πω πως ε, μία πρώτη ανάλυση δική μας λέει πως ε, θεωρώ πως πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο λεπτομερώς και το να πούμε ναι ή όχι νομίζω πως ε, δεν είναι σωστό για τέτοιου είδους προτάσεις και ενδιαφέρον είναι να ακούμε πως ε, η πιθανή αξία είναι 500 δισεκατομμύρια λίρες για τις βρετανικές ασφαλιστικές εταιρείες σε κάποιο βάθος χρόνου. Εμένα δεν μου έδωσαν τέτοιο νούμερο οι Γερμανοί, οπότε δεν το χρησιμοποιώ. Ε, αλλά ε, πράγματι η νομοθεσία αυτή είναι πολύ σημαντική. Άρα γνωρίζουμε πως ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη νευρικότητα και πρέπει να πω πως δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το ότι δεν είδαμε τα εκτιμώντας, είδαμε μόνο το διατακτικό. Οπότε, εγώ έκανα μερικά τηλεφωνήματα και διαπίστωσα πως ε, τα εκτιμώντας είναι γνωστά, είναι γνωστά στον κλάδο, είναι γνωστά στις εθνικές αρχές. Εμείς γιατί δεν τα έχουμε. Εγώ θέλω ολόκληρο το πακέτο. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Ειδικά όταν ακούω πως ε, περιέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες, παραδείγματο χάρη, όταν μιλάμε για τα ασφάλιστρα. Ένα από τα εκτιμώντας τονίζει πως αυτό ισχύει και για τα ομόλογα ε, και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Επίσης τα εφαρμοστικά μέτρα δεν καλύπτουν όλες τις ε, δυνατότητες ε, της οδηγίας περιφερικιότητας 2, η οποία όπως ξέρετε είχε ορισμένα πρέπει και ορισμένα ίσως. Στα πρέπει όλα είναι καλά. Στα ίσως Εκεί όπου υπήρχε η δυνατότητα εφαρμοστικών διατάξεων χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα από αυτά και υπάρχουν 7 τα οποία δεν ε, εφαρμόστηκαν. Μιλάμε δηλαδή για μια προσέγγιση ήπια, μη υποχρεωτική. Οπότε αναρωτιέμαι γιατί δεν καλύψατε όλα τα ίσως. Ε, και μπορώ να μπω και σε λεπτομέρειες, γιατί νομίζω πως έχουν πολιτική σημασία. Είναι σημαντικό να μην πούμε απλώς ναι όλα καλά γιατί αν δεν καλυφθεί τώρα κάτι στις εφαρμοστικές διατάξεις μπορεί εμείς ε, να πούμε ως κοινοβούλιο πως θέλουμε να καλύψουμε κάποια από αυτά τα ζητήματα με τις δικές μας αρμοδιότητες. Τώρα το ζήτημα όλων αυτών των ασφαλίστρων. Εκεί πέρα πρέπει να πω πως ξέρετε τη θέση μας ε, Συμφωνώ με τον Μπουρκχαρτ πως ε, για τα μάτσιν αυτά τα ασφάλιστα δεν υπάρχει πολύ ισχυρή αιτιολόγηση αλλά και τα αντικυκλικά ασφάλιστα εκεί πέρα υπάρχουν κάποια προβλήματα λογικής πρώτα απ' όλα λοιπόν υπάρχει ασφάλιστο εάν ε, πέσουν ε, πάρα πολύ τα χρηματιστήρια και οι υπόλοιπε χρηματαγορές αλλά Εάν ε, ανέβουν πάρα πολύ, τι συμβαίνει τότε. Γιατί δεν υπάρχει τότε αποζημίωση για κάτι τέτοιο. Ε, αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Ε, δηλαδή ζήτημα συμμετρίας, αν θεωρούμε πως χρηματαγορές υπερβάλλουν, μπορούν να υπερβάλλουν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Γιατί καλύπτεται μόνο η μία κατεύθυνση. Το δεύτερο ερώτημα, για να το θέσω στην Επιτροπή σας σύντομα. Δεν ξέρουμε, και αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα, ε, τι είναι η υπερβολή και τι είναι η πραγματικότητα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι θα είχε συμβεί αν είχαμε αντικυκλικό ασφάλιστρο στα ομόλογα της ελληνικής κυβέρνησης. Θα ήταν αυτό προφύλαξη για τους ασφαλισμένους. Δεν νομίζω. Οπότε θεωρώ πως υπάρχει ένα πρόβλημα και αν θέλετε να καλυφθεί αυτό το ζήτημα της υπερβολής και καταλαβαίνω πως απασχολεί τον κλάδο και αυτό το οποίο είπε η Σάρον την προηγούμενη φορά πως αυτό δεν απασχολεί μόνο τον κλάδο αλλά και τους ασφαλισμένους αν είναι να έχουμε τέτοια προσέγγιση νομίζω πως όπως προτείναμε Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε λοιπόν δεν είναι ασφάλιστρο, αλλά κάποιες ε, προφυλάξεις. Εάν λοιπόν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στις αγορές, θα πρέπει να υπάρχει προφυλάξεις και προς τις δύο κατευθύνσεις και όχι ένα δώρο προς τον κλάδο, ένα ασφάλιστρο δηλαδή. Και συμφωνώ πλήρως με την παρατήρηση του Μπουρκχαρτ πως δεν έχει δοκιμαστεί τίποτα. Δηλαδή να έχουμε τόσο εκτεταμένα μέτρα χωρίς να γίνουν έλεγχοι. Εσείς συνήθως επιμένετε και ε, μου κάνει εντύπωση το ότι εδώ πέρα δεν έχετε πρόβλημα. Γιατί έχουν εντύπωση πως ε, ζητάτε πάντα να γίνεται έλεγχος ε, όταν ε, συμβοδίζει αυτό με τα συμφέροντά σας. Δεν είναι αστείο, γιατί πράγματι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο κλάδος και κρατάει κεφάλαια μακροπρόθεσμα. Οπότε, εάν είναι να εισαχθούν τόσο σημαντικά μέτρα, δεν θα πρέπει απλά να ακούμε κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και να έχουμε ειδικά εκτι, ε, εκτιμώντας για λογαριασμό της Generali στην Ιταλία, γιατί ανησυχούν για τα κρατικά ομόλογα. Βεβαίως, σε μια κατάσταση στην οποία ξέρουμε πως πολλοί επενδυτές αμφισβητούν την ικανότητα κάποιων κρατών μελών να αποπληρώσουν το χρέος τους. Και τι θα συμβεί αν πράγματι δεν μπορούν να αποπληρώσουν το χρέος του. και υπάρχει αυτό το ασφάλιστρο. Έχουμε μετά ζητήματα φερεγγιότητα. Εγώ θα ήθελα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ε, να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με τη σταθερότητα του κλάδου και να πάρουμε σοβαρά το ποια μέτρα θα λάβουμε και θα ήθελα να επισημάνω πως στις εφαρμοστικές διατάξεις υπάρχουν και άλλα προβλήματα όπου δεν λάβουμε υπόψη την ε, άποψη του ΣΕΟΠΣ και ε, υπάρχουν ασθενέστερες προτάσεις. Προφανώς υπό την πίεση του κλάδου. Αυτό καλύπτει ζητήματα όπως η ρύθμιση των κινδύνων μετοχών και spread. Εκεί πέρα στο άρθρο 115 τονίζεται τα ζητήματα μετοχικού κεφαλαίου 39% της ε, αξίας αγοράς. Το ΣΕΟΠΣ είχε προτείνει 45%. Παρόμοιο ζήτημα με στρατηγικές ε, συμμετοχές, ε, το ζήτημα αλωτών αναταραχών όπου της κινητικότητας της αγοράς όπου επίσης δεν ελήφθη υπόψη ο και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα των προσδοκόμενων κερδών και των ιδίων κεφαλαίων. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Νομίζω πως οι εφαρμοστικές αυτές διατάξεις είναι ζητήματα στα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε μόνο με ένα ναι ή με ένα όχι. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω του συναδέλφους να έχουμε μια δημοκρατική συζήτηση και να δοθεί δυνατότητα να ξανανοίξουν οι ε, τροπολογίες. Γιατί για μένα τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς τροπολογίες. Και δεν ήταν δυνατόν να υποβάλουμε τροπολογίες καθώς δεν ξέραμε τα εφαρμοστικά αυτά μέτρα. Οπότε, αναμένω τις συζητήσεις. Και Δεδομένης της ε, κατάστασης κάποιων ασφαλιστικών εταιριών με τα χαμηλά επιτόκια αυτή τη στιγμή, θεωρώ πώ υπάρχει σοβαρή δουλειά που πρέπει να γίνει και αναμένω τι συζητήσει που θα γίνουν. Κάτι άλλο να αναφέρω. Ε, αναμένω την άποψή σας για τις ε, τροπολογίες μας για την αξιολόγηση, γιατί υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα που δεν έχουμε καλύψει και κάνουμε κάποιες προτάσεις για να μην βασιζόμαστε υπερβολικά στις αξιολογήσεις στον τομέα των ασφαλιών και θα ήθελα να ακούσω την άποψη των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το τεράστιο έργο που έκανε αναζητώντας συμβιβαστικές λύσεις. Θα ήθελα να επισημάνω ένα δευτερεύον θέμα, αλλά εξίσου σημαντικό, σχετικά με την τριμηνία αναφορά. Χαίρομαι που η ECR για μία φορά συμφωνεί με την απόφασή μου ε, και συνήθως δεν συμφωνούμε εμείς ως σοσιαλιστική ομάδα. Είμαι βέβαιη όμως ότι θα βρεθεί λύση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να εισαγάγουμε νομοθεσία επίπεδου 1 με βάση ένα αυθαίρετο κατόφλι. Δεν ξέρω πώς καθορίζεται το κατόφλι, αλλά πάντως ρώτησα νομικούς ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και εντυπωσιάστηκα μαθαίνοντας ότι το 99% δεν θα καλύπτεται από τις αναφορές. Άρα λοιπόν τι νόημα έχει η νομοθεσία. Και βέβαια δεν νομίζω ότι αυτό ήταν ο στόχος σας όταν καταθέσατε την πρόταση. Ελπίζω λοιπόν ότι αν καθορίσουμε ένα αυθαίρετο κατόφλι δεν θα βοηθήσουμε από την άλλη να υπάρξει ανεξέλεκτο πεδίο. Και αν οι προδιαγραφές αυτές δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, τότε θα εισαχθούν αυθαίρετα από τους, τις ρυθμιστικές αρχές. Και άρα αυτό ξαναθέτει το θέμα της αναφοράς. Πρέπει να αναζητήσουμε μια λύση, γιατί συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θέλουμε να έχουμε επιπλέον βάρος και φόρτος της επιχείρησης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διαρωτηθούμε τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, θα πρέπει οι προδιαγραφές να εφαρμόζονται αναλογικά ή να προσφέρονται, ας πούμε, δωρεάν, γιατί το βασικό θέμα είναι να μειωθεί το βάρος πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να αναζητήσουμε λοιπόν λύση αλλά όχι με, μια, με ένα αυθαίρετο κατόφλι. Δεν νομίζω όμως ότι είναι σωστό να αναφέρουμε αριθμούς, τιμές, διότι οι τιμές δεν μπορούν να σταθούν σε μια νομοθεσία. Χρειάζεται ε, ε, συνεχή αναθεώρηση τιμών κλπ. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς πρέπει να περιλάβουμε στην νομοθεσία θα πρέπει να είναι ένα σύστημα και όχι συγκεκριμένες τιμές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Νομίζω ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει λίγο από τότε που ε, υιοθετήσαμε την Οδηγία Περιφερεγγιότητας 2. Δηλαδή, ε, πρέπει να εξετάσουμε ε, πολύ σοβαρά τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων που λαμβάνουμε όσον αφορά τα ασφάλιστρα, τις επιπτώσεις, τις χρηματοοικονομικές αγορές κλπ. Να βρεθεί δηλαδή αυτή η ισορροπία μεταξύ ε, ρυθμίσεων και διαφάνειας, ούτως ώστε να μην φορτώνουμε τις, επιχειρήσεις με επιπλέον βάρος. Από την άλλη, οι επόπτες θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες. Η οδηγία Φερεγγιότητα 2 ε, ήταν αυτή που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό αυτό που συνέβη ε, με τα ομόλογα και ιδιαίτερα με τα κρατικά ομόλογα. Συμφωνώ με τον Φεν ότι όταν μιλούμε για ε, κυκλικά buffers, κυκλικά ε, προστατευτικά, αυτά μπορούν να βοηθήσουν, αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ασφαλιστικά ταμεία ε, βεβαίως απόλαυσαν τα ωφέλη των καλών εποχών, αλλά δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει κανείς να λάβει υπόψη το χρόνο και όταν η αγορά πέφτει αυτό επιδεινώνει τα πράγματα. Βεβαίως. Θα πρέπει να περιλάβουμε τα, ε, κρατικό χρέος ε, στο οδηγία Φερενγκιότητα 2 να πω δύο πράγματα σχετικά με την ανάθεση ε, δράσεων ή ενεργειών, για να μην παρέμβω ως πρόεδρος κάθε φορά. Δεν νομίζω ότι σκεφτήκαμε παρκώς ή λάβαμε υπόψη όλες τις συνθήκες όσον αφορά το ε, χρονοδιάγραμμα, το περιθώριο χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας. Όταν κάναμε την λισαβονοποίηση, Lisbonization, δεν λάβαμε υπόψη τα τεχνικά standards και τα χρονικά περιθώρια που απαιτούνται υπό διάφορες συνθήκες με βάση τη νέα οδηγία. Το εφεύραμε αυτό στο πλαίσιο της υπάρχουσας οδηγίας με κάποιες μικρές αλλαγές. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ένα εντελώς νέο ε, πεδίο με ένα εντελώς νέο κείμενο. Άρα λοιπόν το ένα συν ένα δεν είναι δυνατό για ένα κοινοβούλιο. Και δεν είναι ε, σωστό να απορρίψουμε κάτι απλώς επειδή δεν είχαμε το χρόνο να το εξετάσουμε ή να δεχθούμε κάτι χωρίς να γνωρίζουμε όλες τις συνέπειες. Άρα λοιπόν, αν έχουμε επαρκή χρόνο να εξετάσουμε σε βάθος τους μηχανισμούς και νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνος πρακτικός τρόπος να προχωρήσουμε. Ε, είπαμε ότι ε, είπαμε ότι θα κάνουμε διότι ξέραμε ότι κάτι μπορεί να γίνει όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη shall, ενώ όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη may, αυτό εισάγει την έννοια της δυνητικότητας. Η Αν υπάρχει χρόνος και υπάρξει δοκιμή, αυτό ισχύει. Όταν λέμε λοιπόν shall ή may υπάρχει διαφορά κάποια από τα ΜΕΙ, ότι θα κάποιες μάλλον από τις ε, φράσεις που χρησιμοποιούμε με τον όρο ΜΕΙ θα πρέπει να αλλάξουν λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα, κατά την εφαρμογή των μέτρων, Σβέν, δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τις, τα εφαρμοστικά μέτρα. Εμείς βέβαια θα καταθέσουμε τις τροπολογίες που θέλουμε και αν ε, υιοθετηθούν, εντάξει. Και νομίζω ότι αυτό έγινε με επιτυχία κατά την προηγούμενη θητεία. Αυτό έγινε και στα εφαρμοστικά μέτρα της MIFID. Δηλαδή έχουμε έναν τρόπο να προωθήσουμε τροπολογίες. Δηλαδή ο Πίτερ θα μπορούσε να εισαγάγει ένα κείμενο με προτάσεις αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ μην θορυβείτε. Η συζήτηση συνεχίζεται για το Omnibus 2. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα απαντήσω σε κάποια από τα σχόλια που έγιναν σήμερα το πρωί πολύ σύντομα. Σχετικά με τη ρήτρα Sunshine εφαρμόζουμε τα μέτρα υπομορφήν πακέτου. Αυτό είναι σημαντικό, διότι υπάρχει ανησυχία στο κλάδο. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν ε, μέχρι πότε θα εφαρμόζεται η οδηγία φερεγγιότητα 2. Και είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί ένας ρυθμός μεταρρυθμίσεων επαρκής για την προσαρμογή. Ε, δεδομένου ότι πρέπει να λειτουργήσει η αγορά σε περίοδο κρίσης. Τώρα, ως προς τις εγγύσεις. Αυτό σχεδιάστηκε ως πακέτο, όπως σας είπα, για να αντιμετωπίσουμε τις ποικίλε καταστάσεις που ισχύουν στις χώρες μέλη, όπου υπάρχουν διάφορα προϊόντα. Γνωρίζουμε και την πτυχή της ανταγωνιστικότητας και τη λαμβάνουμε υπόψη. Άρα, λοιπόν, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι επαρκώς διαφανή. Γι' αυτό λοιπόν στα εφαρμοστικά μέτρα του σχεδίου έχουμε λάβει υπόψη την πτυχή της διαφάνειας. Η πτυχή της αναφοράς είναι πολύ σημαντική. Η φερεγγιότητα 2 δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την απαραίτητη, το απαραίτητο σύστημα αναφοράς. Άρα λοιπόν οι επόπτες έχουν ανάγκη των δεδομένων για να μπορέσουν να εποπτεύουν την αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν καλύτερο να αναζητηθούν λύσεις με βάση την πραγματικότητα και να περάσει και αυτό το μήνυμα στους επόπτες. Ετέθη το ερώτημα σχετικά με την sovereigns, λέει ο μιλητής, ε, υπό την οδηγία φερεγγιότητα 2 έχουμε μία αρχή ε, μια αρχή που αφορά τη μία αγορά ως προς την άλλη. Αυτό βοηθά τον κλάδο και ως ένα βαθμό έχουμε λάβει υπόψη αυτό το ε, στοιχείο. Ως προς τα σκεπτικά. Γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη. Απαντώ. Αυτό είναι απλώς ένα σχέδιο, δεν είναι το πακέτο το οριστικό. Γι' αυτό λοιπόν δεν διανεμήθηκαν τα σκεπτικά και δεν διανεμήθηκαν ούτε στις χώρες μέλη, ούτε σε κανέναν άλλον, διότι βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι ε, της επεξεργασίας. Τώρα, ως προς τα εφαρμοστικά μέτρα. Συμφωνώ μαζί σας. Όταν υιοθετήθηκε η οδηγία πλαίσιο, υπήρχε, υπήρχε ο όρος May. Ε, τότε διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με αυτή την ε, διατύπωση, γιατί σε πολλούς τομείς χρειαζόταν μεγαλύτερη εμπειρία. Τώρα, ως προς τα κυκλικά ασφάλιστρα. Αυτή τη στιγμή σε πολλούς τομείς υπάρχουν προστατευτικά μέτρα, κάποιες φορές και καλυμμένα. Εμάς στόχος μας είναι τα πάντα να είναι διαφανή. Αλλά σε περιόδους κρίσης είναι σημαντικό τα αντικυκλικά μέτρα να αποτρέπουν την, ε, τις διακυμάνσεις, διακυμάνσεις οι οποίες δεν βοηθούν καθόλου την αγορά. Το matching premium είναι ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζεται σε πολύ ειδικέ συνθήκες, όπου δηλαδή ε, το ασφάλιστρο θα είναι αρνητικό στις καλές εποχές και θετικό στις κακές εποχές. Αυτό, κυρία Πρόεδρε, ως ε, αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα όσα συζητούμε. Ο Μπέρκαρτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζω τον περιορισμό του χρόνου και ξέρω ότι έχουμε ψηφοφορία. Θα είμαι πολύ γρήγορο στα σχόλια. Δύο πράγματα. Στον Πίτερ Σκίνερ. Ο Πίτερ Σκίνερ είπε ότι κατά την άποψή του το matching premium είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν είμαι απόλυτα ε, βέβαιος επ' αυτού. Ε, σχετικά με τις μικρομεσαίες. Πράγματι, πρέπει να υπάρξει ειδική μεταχείριση στο πλαίσιο αυτό και πρέπει να αναζητήσουμε μία απάντηση. Σιντεγκούλα είπε να μην ξεχάσουμε τον ανταγωνισμό όταν μιλούμε για ασφάλιστρα. Πράγματι, έτσι είναι. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα, υπάρξει, θα υπάρχει εναρμόνιση και από την πρώτη στιγμή, το σημείο εκκίνησης. Γι' αυτό το 1, 3 και 8 ε, αυτό ακριβώς επιδιώκουν. Ε, υπάρχει ε, ορθή νομική βάση επ' αυτού. Ένα άλλο σχόλιο έλεγε ε, δεν θα πρέπει να υπάρχουν, να θεσπιστούν κριτήρια για το πότε και πώς ε, η ΑΙΟΠΑ δηλώνει κατάρρευση συστήματος. Ναι, βεβαίως, ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτό επιδιώκουμε εδώ και, και καιρό. Ε, πράγματι όπως σχολιάστηκε πρόκειται για ένα πολύ ογκώδες πακέτο και, το, και βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα χρονοδιαγράμματα μέσα στα οποία λειτουργούμε. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σήμερα το απόγευμα όταν θα υπάρξει μια συνάντηση μεταξύ των σκιωδών. Ο Σφέν Κίγκολ ε, ρώτησε για ποιο λόγο δεν λάβαμε ακόμα τα σκεπτικά. Ε, την περασμένη εβδομάδα επικοινώνησα με την ε, Επιτροπή και μάλιστα και με τον ίδιο τον Μισελ Μπαρνιέ ζητώντας ακριβώς το λόγο. Πριν ολοκληρωθεί η έκθεση νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και το σκέλος του σκεπτικού από πλευράς ε, κομισιών. Στην κυρία Μακάρθη. Νομίζω ότι τα σχόλια αυτά έχουν ληφθεί υπόψη και θα βρούμε ε, λύση. Ε, επ' αυτού. Δηλαδή, ε, εκεί στο σημείο όπου δίδονται τιμές ή ποσά, ε, αυτά θα αντικατασταθούν με κάποιες, με περιγραφή μηχανισμού. Έρχομαι τώρα στο δικό σας σχόλιο τείνω να συμφωνήσω μαζί σας κυρία Πρόεδρε. Ασφαλώς θα απαιτηθεί χρόνος για να υπάρξει δικαιοσύνη. Και να μην ξεχνούμε ότι ο βασικός στόχος της έκθεσης αυτής είναι να επιδιωχθεί μια ισορροπία. Ακριβώς αναζητείται αυτή η ισορροπία. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους οι οποίοι με βοήθησαν πραγματικά στο έργο μου και σήμερα το απόγευμα στις 5 θα έχουμε μια συνάντηση του εισηγητή με τους σκιώδεις και νομίζω ότι για πολλούς από εμά αυτό ε, ε, θα είναι πολύ αποτελεσματικό. Η Πρόεδρος. Και τώρα στις 19 και 20 Δεκεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία ώστε να φτάσουμε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Καθυστερήσαμε λίγο γιατί έπρεπε να περιμένουμε κάποια μέλη. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να κερδίσουμε χρόνο για να δούμε αν μπορούμε να το πράξουμε αυτό. Πάμε στο 5 που είναι η ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να είμαστε όλοι έτοιμοι για την ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις κάρτες σας, τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Καταρχήν, θα ήθελα να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Okay, with two socialist cards down anymore. Δύο σοσιαλιστές μείον. Μπορείτε σας παρακαλώ να πατήσετε τα κουμπιά σας. Yeah, I We've got 39 cards. that... 39 κάρτες έχουμε και έχουμε δύο λιγότερους σοσιαλιστές. Υπάρχουν άλλα προβλήματα. Δύο δεν ε, πίεσαν το κουμπί τους. Τώρα έχουμε έναν επιπλέον από τους φιλελεύθερους. Ωραία, δεν θα ψηφίσω εγώ τότε. Μου διευκολύνεται το έργο. Κάποιος δεν έχει πιέσει το κουμπί. Ε, ελέγχω για να δω κατά πόσο φταίει το δάχτυλό σας ή η μηχανή. Α, εσείς ήσασταν. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα. Έχουμε δύο σοσιαλιστές λιγότερους, όπως είπα. Συμβασμός Α, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω. Ήμκο 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 13 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε. Σας παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία για ΙΜΚΟ 13. Everybody... Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 4 was carried. Ίμκο 4 πέρασε. Θέλετε να ελέγξουμε το ΙΜΚΟ 4. ΙΜΚΟ 4 ελέγχουμε ηλεκτρονική, η οποία και αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίθηκε 27 υπέρ, 11 κατά. Σίγουρα εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Β σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Έκτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έβδομο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όγδο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σας προειδοποιώ ότι δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο έκτο, ε, οκτώ τμήματα σε ένα συμβιβασμό. 16 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα το ελέγξω εφόσον το επιθυμείτε. Ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ και 18 κατά. Συμβασμός Δέλτα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σε ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Compromise F in τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά απο... αποχές απορρίπτεται. 41 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός G, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Με συγχωρείτε, παράγραφος 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ ε, κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα μεταξύ των υπέρ και των αποχών. Ψηφίσατε όλοι 52. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίφθηκε. H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 8 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ ΙΜΚΟ 8 ελέγχουμε ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίφθηκε 58 υπέρ κατά αποχές ε, μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ αρχίζει η ψηφοφορία για την 58 ψηφίσατε όλοι πέρας Πώς πρόσθετους επιπλέον έχουμε από τους σοσιαλιστές 2, άρα 21 κατά 20 υπέρ, άρα ε, απορρίπτεται. Ήμκο 14 Α, έκανα λάθος. Οι σοσιαλιστές ψήφισαν υπέρ. Δεν καταψήφισα. Άρα 20 συν 2. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει η ΜΚΟ 14 σε αυτή την περίπτωση. Δεν έχω ελέγξει πόσοι είναι οι σοσιαλιστές. Πρέπει να έχετε τις κάρτες σας στο μέλλον παρακαλώ. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα ήθελα να ελέγξουμε την 60 αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται γιατί οι σοσιαλιστές αυτές. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Α, συμβιβασμό υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο τμήματα, 63 πρώτο μέρος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 64 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 66 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, μπορούμε να ελέγξουμε την 66 παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήμκο 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Μπορούμε να ελέγξουμε την 73 παρακαλώ. Αρχίζει η ηλεκτρονική Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Ήμκο 9 υπέρ. Κατά. Σας παρακαλώ πάλι. Ήμκο 9 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Ήμκο 11 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ. Δεν είναι σαφές. Μου λείπουν μερικοί από ορισμένε ομάδες. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Είσαστε υπέρ. Εγκρίνεται. 74 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μα εννοούσα τρία. Τραν τέσσερα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν πέντε. πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν εξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν επτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν οκτώ υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρη γιατί δεν βλέπω ότι κάνετε μερικοί. Ελέγχουμε. groups put their hand up, I can't tell. Δεν είμαι σίγουρη για ορισμένες ομάδες. Πέρας και απορρίπτεται. Τραν 9, πρώτο τμήμα, υπέρ. Μεταφορές 9, πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τραν 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τραν 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 21, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, θέλω να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 21. Νομίζω πέρασε αλλά δεν είμαι σίγουρη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Με έναν σοσιαλιστή επιπλέον. 22 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10, 76 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικέ σκέψει 11 με 19 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά επί του κειμένου όπω έχει τροποποιηθεί. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. 39 υπέρ, 40 μάλλον, 42 κατά και καμία αποχή. Άρα να συγχαρούμε τον ε, εισηγητή. Θέλει ο εισηγητής να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την στήριξη και την ε, καλή συνεργασία με τους κοιόδες εισηγητές. Να αναφέρω κάτι με ευκαιρία την 40η επέτειο της έκθεσης ε, φέτος ε, επικεντρωθήκαμε σε ορισμένα ε, ζητήματα και κάποιες τροπολογίες δεν μπόρεσαν να ενσωματωθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτονται, απλά μόνο ότι επικεντρωθήκαμε σε ορισμένα ζητήματα. Αυτό ήθελα μόνο να προσθέσω. Ευχαριστώ. Uh, I'm very sorry I was being... Λεπάμε. Συγχωρείτε με ενημέρωναν. με ενημέρωναν, οπότε δεν άκουσα τι είπατε. Κάποιο θα μου το πει μετά. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα έχουμε άλλο ένα θέμα, ψήφιση της ε, προφορικής ερώτησης για το σχέδιο πίνακα βαθμολογίες. Νομίζω πως οι πρώτες 7 ερωτήσεις μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Πρώτες 7 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. Ερώτηση 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κείμενο της έδρας της έκτης ερώτησης. Ψήφισαν όλοι. Συνεχίστε να ψηφίζετε. Πατήστε τα κουμπιά. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Όχι, όχι, μην, το, μην βγάζετε την κάρτα. Κάποιοι έβγαλαν τις κάρτες πριν ε, τα αποτελέσματα. Ξαναβάλτε τις. Ωραία, πέρας. 39 υπέρ. Ωραία. Τα γελία πράγματα ψηφίζουν και φεύγουν. So,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 Okay, those who are not staying, please uh, leave the room quietly. Λοιπόν, ε, όσοι δεν θέλουν να μείνουν στην αίθουσα, παρακαλώ να φύγουν ήσυχα. Περνάμε στο σημείο 6. Ε, θέση για κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για την έκδοση κερμάτων ευρώ. Τον λόγο έχει ο εισηγητής ο Χάνς Πέτερ Μάρτιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Ε, βλέπετε, φύγαν οι συνάδελφοι για μεσημεριανό διάλειμμα. Ευχαριστώ για τις τροπολογίες. Μιλάμε κατ' ουσίαν για τις τροπολογίες των συναδέλφων από την Ουγγαρία. Πρώτα έχουμε την υπαριθμόν 14, όπου μιλάμε για θρησκευτικά ζητήματα τα οποία τα σχέδια δεν πρέπει να προσβάλλουν ούτε να φύγουν θρησκευτικού προσανατολισμού άλλων κρατών μελών. Ε, αυτό προτείνω να ευθυγραμμιστεί με την τροπολογία και προτείνω το κείμενο το οποίο σας είπα. Τα σχέδια δεν πρέπει να προσβάλλουν ε, θρησκευτικούς ή άλλους προσανατολισμούς ε, και πεπιθήσεις. Οπότε καλύπτεται νομίζω έτσι. Ε, υπάρχουν και άλλες τροπολογίες από τους συναδέλφους στους οποίους, οποίους υποστηρίζω. Οπότε νομίζω πως με βάση τις συζητήσεις με την Κομισιόν προετοίμασα άλλες τρεις τροπολογίες και θα γίνει μια προσπάθεια να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο στο σχεδιασμό των νομισμάτων. Ε, δεν εννοώ ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να υπάρξει ίσως, δεν ξέρω, μια συμμετοχή κάποιων συναδέλφων ε, ή ο πρόεδρος ε, είτε ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ε, να μείνει με αυτόν τον τρόπο στην ιστορία εάν επιλέξει το επιτυχημένο σχέδιο. Το επόμενο ζήτημα, μια επιθυμία, προθεσμία για τιμητικά νομίσματα διαφόρων επαιτίων να μειωθεί και από δύο χρόνια να γίνει έξι μήνες. και αυτή την υποστηρίζω και μετά υπήρχε και άλλη μια επιθυμία την οποία αντιλαμβάνομαι να μην καλύψουμε μόνο τα κανονικά νομίσματα αλλά και τα συλλεκτικά ε, όσον αφορά το θέμα της προσβολής ε, θρησκευτικών ε, πεπιθήσεων και λοιπόν πεπιθήσεων τέταρτων και συναρπαστικό, αν θέλετε, η επιθυμία μας να εισαχθούν χαρτονομίσματα του ενός και των δύο ευρώ. Παρά το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Συμβούλιο δεν το θέλουν. Εγώ θα επιμείνω και θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε πως η Κομισιόν πρέπει να ερευνήσει το ζήτημα αυτό τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά είχαμε μια τοποθέτηση από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Οπότε αυτό θα τεθεί ως αίτημα, όχι ως τροπολογία. Νομίζω πως έτσι θα γίνει και πιο ζωντανή συζήτηση. Ευχαριστώ. Μάλιστα, είμαστε στα σημεία 6 και 7 μαζί, αν είχατε κάποια αμφιβολία. Ζαν Πολ, θέλετε να παρεμβείτε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή για την εργασία του για αυτές τις δύο εκθέσεις οι οποίες ε, δεν είναι τόσο μεγάλες σε όγκο, αλλά αφορούν όλους τους Ευρωπαίους. Αν υπάρχει ένα ε, στοιχείο που αφορά 17 χώρες, είναι τα κέρματα ευρώ. Και όπως είπα την ε, προηγούμενη φορά, υποστηρίζω την ιδέα ότι μας χρειάζεται το νόμισμα του ενός ευρώ Ξέρω ποια είναι τα σχόλια της ΕΚΤ για το κόστος νομίσματοκοπής, αλλά νομίζω ότι έχει συμβολικό χαρακτήρα και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται. Ναι, να δίνουμε φιλοδορήματα σε ευρώ αντί για δολάρια. Ε, ε, ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες αυτές τις προτάσεις. για τα χαρτονομίσματα τώρα ενός και δύο ευρώ. Ο δεν μπορώ να το στηρίξω για το λόγο που αναφέρθηκε Μιλάμε για την έκδοση κερμάτων εδώ πέρα. Δεν είναι νομίζω το σωστό σημείο για αυτή την πρόταση. Αλλά βεβαίω. Εντάξει. Αφήστε που εγώ δεν βλέπω και την ανάγκη για κάτι τέτοιο. Νομίζω πως ε, όσον αφορά δε το σχεδιασμό των νομισμάτων εγώ θεωρώ πως πρέπει να εξακολουθήσει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και τέλος δεν υποστηρίζω τις σχετικές τροπολογίες. για το πώς πρέπει να κυκλοφορούν τα νομίσματα του ενός και των δύο ευρώ. Ευχαριστώ, Σόφη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξέτασα με ενδιαφέρον την έκθεση του κυρίου Μάρτιν. Κάποιες προτάσεις δεν θα μπορέσουμε να τις στηρίξουμε όσον αφορά τα χαρτονομίσματα ενός και δύο ευρώ. Μήπως θα ήταν καλό να το συμπεριλα... να συμπεριλάβουμε ε, τις ε, τροπολογίες Τρεμόζα που ζητάει αξιολόγηση της ε, έκδοσης ε, νομισμάτων ε, ενός και δύο λεπτών και να αξιολογήσουμε συνολικά το ζήτημα και για τα χαρτονομίσματα ενός και δύο ευρώ. Ένα γενικότερο για το σχέδιο των νομισμάτων σε κάποιες από τις προτάσεις του εισηγητή αλλά και σε κάποιες τροπολογίες έχω την αίσθηση πως μπορεί το ζήτημα αυτό να οδηγήσει σε κάποιες ε, συγκρούσεις. Αν έχουμε ενιαίο νόμισμα, πρέπει να είναι κάτι το οποίο μας ενώνει. Και θα είναι λυπηρό να γίνει εθνικιστικό ζήτημα. Η ζήτημα θρησκείας. Αν έχουμε ένα κοινό νόμισμα, πρέπει να μας ενώνει. Και όχι ζήτημα του τι προσβάλλει την άλλη χώρα ή την άλλη θρησκεία. Οπότε τελικά επαφίεται στα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να φροντίσουν να είναι αποδεκτά τα σχέδιά τους. Κανείς άλλος δεν θέλει να μιλήσει, από τον λόγο έχει πάλι ο Χάνς Πέτερ. Ναι, σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Όσον αφορά τα χαρτονομίσματα, να υπενθυμίσω πως στους τροπολογίες μου λέμε απλά να θέσουμε το ζήτημα. Τίποτα άλλο. Τώρα ε, είναι λυπηρό οι σοσιαλδημοκράτες για τεχνικούς λόγους να εμποδίσουν αυτή τη συζήτηση. Το έχω πει νομίζω πολλές φορές. Είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε το τι ε, εικόνα δίνουμε ειδικά σε καιρούς Κρίση. Υπάρχουν υπέρ και κατά, αλλά νομίζω πως υπάρχει μια πλειοψηφία εντός του Κοινοβουλίου για, να... για το ζήτημα αυτό. Νομίζω μπορεί να ξαναξεκινήσει η συζήτηση. όσον αφορά την κυρία Ενετφέλτ πράγματι αυτό που λέτε είναι λογικό με την αξιολόγηση των ε, κερμάτων του ενός και δύο λεπτών να αξιολογήσουμε και τα χαρτονομίσματα του ενός και δύο ευρώ και προσωπικά ε, υπάρχει και αυτό το σύστημα, ξέρετε, αυτών των τιμών, τα 14,99 που πολλοί πελάτες θέλουν και το, το, το ένα λεπτό, το ένα σεντ ρέστα. Επίσης, για τι άλλε απολογίες. Είναι λυπηρό να υπάρξει αυτή η ερμηνεία την οποία είχατε κι εσεί. Εγώ θα επιθυμούσα να μην υπάρχει τίποτα το προσβλητικό από μια χώρα προ μια άλλη και ε, τίποτα το θρησκευτικό ακριβώ για να υπάρχει αυτή η, ε, έννοια του ότι μα ενώνει και όχι ότι μα χωρίζει κάτι. Έτσι το, το ερμήνευσα εγώ. Ναι, να σου το πω εγώ θεωρώ πως αν μια χώρα π.χ. έχει αντισημιτικά σύμβολα να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν το θέμε. Αλλά α, δεν είναι τώρα τίποτα άλλο. Να, δεν είναι δουλειά μας να μπούμε στα χωράφια των κρατών μελών και της επικουρικότητας. Νομίζω λοιπόν ότι λογικότερα θα ήταν αυτή η διατύπωση που πρότεινα. Όχι, όχι στο πλαίσιο λοιπόν έτσι, εθνικισμού και να αρχίσει ο ένας να πικάρει τον άλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε στις 29 Νοεμβρίου. Αυτές είναι οι προθέσεις μας και να συζητηθεί στην, ολομέλεια, στην πρώτη Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ όλους. Αυτά ήταν τα θέματα 6 και 7. Λίγουν τα θέματά μας για σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 3 έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο και θα τελειώσουν οι εργασίες μας στις 5. Και στη συνέχεια θα συνεδριάσουν ε, πολλοί σκιώδεις ε, από όσο γνωρίζω. Θα σας δω το απόγευμα στις 3. Γεια σας.